Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε. Και λίγο ησυχία για να ξεκινήσουμε. Yes. Σας ευχαριστώ πολύ όλους που, για την παρουσία σας. Ε, Καλώς ορίσατε. Να καλωσορίσουμε θερμά και τους προσκεκλημένους μας εδώ στο βήμα. Θα τους ανακοινώσω έναν προς έναν αμέσως μετά τα διάφορα διαδικαστικά. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης της έκτακτης συνεδρίασης της Επιτροπής ε, ΛΥΜΠΕ για τις πολιτικές ελευθερίες και την εσωτερική ε, ασφάλεια έκτακτη γιατί είναι πάρα πολύ ε, βεβαρημένη η εβδομάδα στις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε σειρά ακροάσεων και η Επιτροπή Λίμπε είναι τόσο σημαντική και είμαστε επί της ουσίας αρμόδια επιτροπή σε τουλάχιστον τέσσερις ακροάσεις, συνδεδεμένοι σε άλλες δύο και είμαστε και προσκεκλημένοι σε άλλες δύο, επομένω είμαστε ιδιαίτερα απασχολημένοι αυτές τις ε, μέρες, αλλά βρήκαμε ε, και χρόνο για να τίνουμε δίκονο σε αυτό το θέμα το οποίο έθεσε η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ μέσω των συντονιστών της στην διάταξη. Ε, τώρα, το γλωσσικό καθεστώς υπάρχει διερμηνία σε όλες τις επίσημες γλώσσες με εξαίρεση τα μαλτέζικα, τα λετονικά και τα ιρλανδικά. Και ευχαριστούμε για την κατανόησή σας. Τώρα, έγκριση των συστάσεων των συντονιστών. Εγκρίνουμε τις συστάσεις βάσει του άρθρου 214 Υπάρχουν ε, ε, σημειώσεις των συντονιστών, ε, τις οποίες μπορείτε να βρείτε μεταξύ των εγγράφων σας. Εγκρίνονται λοιπόν οι συστάσεις, αν δεν κάνω λάθος, και μπορούμε να περάσουμε στο σημείο που έχουμε σήμερα προς τη συζήτηση, η ακρόαση για την έρευνα και διάσωση στη Μεσόγειο. Είναι ένα θέμα ιδιαίτερα σημαντικό. Παρακαλώ κύριε Μαχίτε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Μία ερώτηση. Μήπως θα τηρήσουμε ετήσια ένα λεπτό σιγής για την ε, ε, επέτειο της λαμπεντούσα Το θυμα... Ναι, ναι, θα το κάνουμε, αλλά αυτό είναι δουλειά του Προέδρου. Θα υπάρχει. Ναι, είναι δουλειά του Προέδρου. Ωραία να περάσουμε στο σημείο αυτό ακριβώς την ημέρησα διάταξη. Ε, κύριε Προκατσίνη, διαδικαστικό. Για να είμαστε βέβαιοι. Θα γίνουν δύο γύροι ερωτήσεων ή μόνο ένας γύρος ερωτήσεων, γιατί δεν κατάλαβα. Ή μάλλον, αν θα μπορεί ο καθένας από εμά να πάρει το λόγο για να διατυπώσει ερωτήσεις δύο φορές ή μόνο μία φορά και αν οι συντονιστέ ε, θα λάβουν το λόγο πρώτοι γιατί δεν ε, ε, το βλέπω αυτό στι σημειώσει. Κύριε Προκατσίνη, περιμένετε λίγο τον πρόεδρο. Περιμένετε τον πρόεδρο της Επιτροπής να, για να ανακοινώσει όχι μόνο το σημείο αυτό στην ημερήσια διάταξη, αλλά και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουμε. Επιτρέψτε μου να συνεχίσω και θα ανακοινώσουμε αμέσως πώς ε, θα διαρθρωθεί η συζήτηση την οποία θα κάνουμε σήμερα το πρωί. Λοιπόν, ανακοίνωνα ακριβώς ε, το σημείο αυτό στην ημερήσια διάταξη. Είναι σήμερα 3 Οκτωβρίου 2019. Είναι εθνική επέτειο στη Γερμανία αλλά είναι και η επέτειος ε, ε ενός ολέθριου γεγονότος, ε, η βήθηση του σκάφους που μετέφερε ε, μετανάστες από τη Λιβύα στην Ιταλία. Πάνω από 360 άνθρωποι χάθηκαν σε αυτό το ναυάγιο το 2013. Πρόκειται για τεράστια τραγωδία και έκτοτε έχουν χαθεί πολύ περισσότερες ζωές και πολλές φορές στην Ολομέλεια, στο Στρασβούργο έχουμε μνημονεύσει αυτές τις τραγωδίες στη Μεσόγειο. Έξι χρόνια λοιπόν μετά από αυτό το σοκ ε, ακόμα χάνονται ζωές ε, στη Μεσόγειο στην προσπάθειά τους ε, να φτάσουν στις ευρωπαϊκές ακτές της Μεσογείου. Το 2016 το Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα ψήφισμα για την κατάσταση στη Μεσόγειο και την ανάγκη, έτσι το αποκαλέσαμε, με μια ολιστική προσέγγισης ε, Δύο αξιότιμα μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ συνυπέγραψαν αυτό το ψήφισμα ω εισηγητές, η κυρία Μέτσολα και ένα συνάδελφο που δεν είναι πλέον εδώ, η Σεσίλ Κιέγγε. για να ε, έχουμε μια νέα προσέγγιση για τη μετανάστευση, για μια πιο εύρωστη και πιο αποτελεσματική απάντηση της Ένωσης ε, στις επιχειρήσεις έρευνας και διάθεσης και να μην έχουμε ε, κλιμάκωση των θανάτων στη Μεσόγειο για τους μετανάστες που προσπαθούν να φτάσουν στις ακτές μας. Το 2018 το Κοινοβούλιο ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει κατευθυντήριες γραμμές ε, για τη λεγόμενη οδηγία διευκόλυνσης προκειμένου να αποφύγουμε την ε, ποινικοποίηση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Μέχρι τούδε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει προτείνει κάτι τέτοιο. Ο ρόλος της Frontex σε αυτές τις επιχειρήσεις έχει ενισχυθεί. Η Uniformed, την ε, επιχείρηση Σόφια, ε, επέκτηνε την εντολή της, αλλά ε, είναι περιορισμένη μόνο σε ε, επιχειρήσεις από αέρος, όχι θαλάσσιες επιχειρήσεις. Και πορικά σκάφη και μη κυβερνητικέ οργανώσεις έχουν γίνει όλο ένα και πιο δραστήρια για την διάσωση ζών στη θάλασσα και θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο και ταυτόχρονα ε, κινδυνεύουν να τιμωρηθούν ενώ ε, προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια. Υπάρχει μια πρόσφατη συμφωνία στη Μάλτα για να ε, υπάρχουν ε, πιο σταθερές λύσεις για την αποβίβαση των ανθρώπων αυτών ε, από τη θάλασσα, αλλά χρειάζεται διευκρινήσεις και πρέπει να διευκρινιστεί και ο ρόλος που πρέπει να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σήμερα λοιπόν έχουμε αποφασίσει να κάνουμε μια ειδική ακρόαση και έχουμε προσκεκλημένους ομιλητές για να μας βοηθήσουν να έχουμε μια σαφέστερη εικόνα της κατάστασης. Να αξιολογήσουμε τι και να υπάρχουν στην νομοθεσία και στις πολιτικές μας και να βρούμε και μία πιθανή άγουσα για το μέλλον. Γι' αυτό ακριβώ και ο στόχος μας είναι να ε, χρησιμοποιήσουμε τη σημερινή ακρόαση για να συντάξουμε στη συνέχεια ένα σχέδιο ψηφίσματος. Ε, θα ψηφιστεί στην Επιτροπή μας ε, στις 21 Οκτωβρίου και θα υποβληθεί στην Ολομέλεια για τη δεύτερη Ολομέλεια του Οκτωβρίου. Στην επόμενη δηλαδή Ολομέλεια στο Στρασβούργο. Θα υπάρχει μια διαδικασία ερωτήσεων και απαντήσεων αφού ακούσουμε τους ομιλητές μας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο Μάικολ Σότερ, ο οποίος θα μας ενημερώσει για τις ε, πρόσφατες εξελίξεις, είναι διευθυντής για τη μετανάστευση, προστασία και θεωρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Τόμας Μόλναρ από το ε, ε, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, τη ΦΡΑ, η κυρία Καρόλα Ρακέτε, η οποία θα μοιραστεί την εμπειρία μας ως ε, κυβερνήτης του Sea Watch που διασώζει μετανάστες στη θάλασσα, τον καπετάνιο Ανδρέα Τασάρα από την Ιταλική Ακτοφυλακή, που θα δώσει την άποψη των Ιταλικών αρχών και τον εκτελεστικό διευθυντή της Frontex, τον Φαμπρίς Λεζερή, ο οποίος θα μιλήσει μαζί μας ε, μέσω σύνδεσης με βίντεο, διότι δεν μπορεί να παρευρεθεί εδώ σήμερα ε, και το αρχηγείο της Frontex βρίσκεται στην ε, Πολωνία, στη Βαρσοβία. Δεν μπορεί λοιπόν να βρίσκεται εδώ όσο συχνά θα θέλαμε, αλλά θα κάνει τις δηλώσεις τους μέσω αυτής της σύνδεσης με βίντεο. Και πριν ε, προχωρήσουμε και να δώσουμε το λόγο στους ομιλητές ε, για 10 λεπτά τον καθένα το πολύ, θα υπάρχουν ε, δύο γύρι ερωτήσεων και απαντήσεων. Σας το επιβεβαιώνω αυτό. Τώρα, να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή εις μνήμην όλων των θυμάτων των τραγωδιών ε, στη Μεσόγειο. Thank ευχαριστώ. Και τώρα προχωρούμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα. Ε, προβλέπεται δύο ώρες συνεδρίωση και έχουμε μέχρι τις 11 λοιπόν. Έχουμε δηλαδή ακόμα 100 λεπτά και πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι πρέπει και οι ερωτήσεις ε, που θα απευθύνετε στους ομιλητές ε, να περιοριστούν στο ένα λεπτό. Ε, έτσι θα μπορέσουμε να δώσουμε το λόγο σε όλα τα μέλη. Θα υπάρχει ένας πρώτος γύρος για τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων και ένας δεύτερος γύρος για όλα τα μέλη που θέλουν να κάνουν ερωτήσεις. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Όπως σας είπα, Πρώτα θα δώσουμε το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, τον Μιχαλ Σότερ, Διευθυντή Μετανάστευσης, Προστασίας και Θεωρήσεων. Έχετε το λόγο για 10 λεπτά το πολύ, παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση σήμερα σε αυτή τη συνεδρία σε ένα πολύ σημαντικό θέμα, την έρευνα και διάσωση στη Μεσόγειο. Η σημερινή ακρόαση της Επιτροπής σας ε, είναι μια ακρόαση που γίνεται σε μια πολύ σημαντική ημερομηνία. Ο αριθμό των θυμάτων έχει πέσει μεν στη Μεσόγειο, παραμένει όμως ακόμα υψηλό και κάθε ζωή που χάνεται είναι και μια τραγωδία. Στις ε, πολιτικές κατευθυντήριε γραμμές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόνισε ότι η διάσωση τη ανθρώπινη ζωής είναι και θα παραμείνει προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι ηθικό καθήκον και υποχρέωση να γίνεται διάσωση ανθρώπων στη θάλασσα και να διώκονται όσοι θέτουν ζωέ σε κίνδυνο. Τώρα πρέπει να βρεθούν τρόποι για μια περισσότερο βιώσιμη, αξιόπιστη και μόνιμη προσέγγιση στην έρευνα και διάσωση και αυτό θα πρέπει να αντικαταστήσει τις προσωρινές λύσεις. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έχουν θεματίσει ρόλο κλειδί στην Μεσόγειο. Έχουν σώσει χιλιάδες ζωές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενίσχυσε τις δυνατότητες διάσωσης στη Μεσόγειο. Τέσσερις επιχειρήσεις έχουν ε, σώσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπινες ζωές από το 2015, 730.000 ανθρώπινες ζωές. Η συμφωνία που βρέθηκε μεταξύ κρατών μελών για την έρευνα και διάσωση δεν είναι τόσο καλή όσο θα έπρεπε και όσο ήταν σε θέματα έρευνας και διάσωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται να κάνει ό,τι μπορεί έτσι ώστε να παρέχει κάθε μέσο για να συνεισφέρει στην διάσωση ανθρώπων στη θάλασσα. Ταυτόχρονα, η πολιτική μας στον χώρο αυτό θα πρέπει να αποτελεί μέρος μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής στον τομέα της ε, μετανάστευσης. Θα πρέπει να είναι συνεκτική, μεταξύ άλλων, με την ε, πολιτική μείωσης ε, των παράτυπων ροών και της ε, δίωξης των ε, διακινητών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει ό,τι μπορεί. Αυτό είπα μόλι. Όμω δεν πρέπει να ξεχνάμε το θέμα τη ε, αρμοδιότητα, διότι είναι μια πολύ σημαντική αφετηρία για κάθε μα δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως γνωρίζετε, η έρευνα και η διάσωση είναι εθνική αρμοδιότητα που ασκείται με βάση το διεθνές δίκαιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, λοιπόν, δεν έχει εξουσία συντονισμού ε, των επιχειρήσεων έρευνα και διάσωση, ούτε μπορεί να ε, ορίζει σημεία αποβίβαση. Αυτό θα πρέπει να γίνει σε συντονισμό με τις εθνικές αρχές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν υπενθυμίζει ότι τα κράτη-μέλη δεσμεύονται από το καθήκον να παρέχουν βοήθεια στα σκάφη που βρίσκονται σε κίνδυνο στη θάλασσα. Αυτό υπαγορεύει το διεθνέ Δίκαιο και το Δίκαιο τη θάλασσα. Υπάρχουν μεγάλες προκλήσεις και σε αυτές πρέπει να ανταποκριθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχοντα στήριξη. Εδώ ήμασταν αρκετά δραστήριοι ε, με διάφορες ε, συντονιστικέ ενέργειες ε, σε τέτοια θέματα. σε 14 περιπτώσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συντονίσει επιχειρήσεις αποβίβασης σκαφών και έχουν ήδη γίνει ενέργειες για την ε, μετακίνηση των μεταναστών στις ε, υπόλοιπες ε, χώρες. Τους τελευταίους δύο μήνες έχουν γίνει επιχειρήσεις και οι διασωθέντες έχουν μπει στη διαδικασία μετεγκατάστασης. Έχουμε λάβει τη στήριξη 15 κρατών μελών και υπάρχει ένας ε, συντονιστικός ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία καταβάλει κάθε προσπάθεια για να δρομολογηθούν οι διαδικασίες μεταγκατάστασης. Ελπίζουμε στο μέλλον, στο προσεχές μέλλον να ξεπεράσουμε τα ε, εμπόδια που έχουν προκύψει σχετικά με το που μπορεί να αποβιβαστεί ένα σκάφος διάσωσης. Στο τέλος Σεπτεμβρίου στη Μάλτα σημειώθηκε κάποια πρόοδο στο θέμα αυτό και το επικροτούμε. Ελπίζουμε και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη να είναι μαζί μας έτσι ώστε να ενισχύσουμε την αλληλεγγύη που οφείλουμε να δείξουμε. Αυτό θα συζητηθεί στο Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων την ερχόμενη εβδομάδα. Ε, παράλληλα θα συνεχίσουμε να παρέχουμε στήριξη και σε επιχειρησιακό και σε ε, πολιτικό και οικονομικό επίπεδο οι διαδικασίες συντονισμού που γίνονται στην Ιταλία και τη Μάλτα αφορούν και τη διαδικασία ασύλου προσπαθώντας να χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένα κριτήρια έτσι ώστε να, διανεμηθεί, να διανεμηθούν οι μετανάστες στα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Παρέχουμε λοιπόν στήριξη μέσω όλων των υπηρεσιών και ευρωπαϊκών οργανισμών, της Frontex μεταξύ άλλων και της Υπηρεσίας Ασύλου. Όμως, σε θέματα έρευνας και διάσωση στη Μεσόγειο πρέπει να αναφερθούμε και στις δραστηριότητες των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λοιπόν, αναγνωρίζει το σημαντικό ρόλο τους στην ε, διάσωση στη θάλασσα και τόνιζε πάντα το πόσο σημαντικό είναι για όλους να ε, διασφαλίζεται η τήρηση του διεθνού ε, δικαίου και, τον, ε, και ο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Χρειάζεται λοιπόν συντονισμό όλων των συμμετεχόντων έτσι ώστε να χαρακτηριστεί με επιτυχία μια επιχείρηση έρευνα και διάσωση. Για το σκοπό αυτό, το 2016, στο πλαίσιο της επιχείρησης Σοφία, ξεκίνησε μια επιχείρηση συντονισμού ακριβώς για αυτό το σκοπό. Σε ό,τι αφορά την ποινικοποίηση τη ε, παροχή ανθρωπιστική βοήθεια σε μετανάστε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει να συνεργάζεται στενά με το Κοινοβούλιο, το οποίο ε, ενέκρινε ένα ψήφισμα σχετικό τον Ιούλιο του 2019. Ποια είναι η ουσία εδώ, ότι καμία ουσιαστική βοήθεια σε μετανάστες που παρέχεται είτε στη θάλασσα είτε σε περιπτώσεις όπου κινδυνεύει η ζωή τους ε, δεν θα πρέπει να ποινικοποιείται. Η αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, στο ευρωπαϊκό πλαίσιο αναγνωρίζει την έλλειψη σαφήνειας ε, του πλαισίου αυτού σε τέτοια θέματα και Αναγνωρίζει επίσης ότι υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω ενέργειες και ε, συνεργασία με τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις έτσι ώστε να ενισχυθούν οι προσπάθειες ε, για την ε, μη ποινικοποίηση των επιχειρήσεων διάσωση. Χρειάζεται λοιπόν να ξεκινήσει ένας διάλογος για την ενδεχόμενη αναθεώρηση των υφιστάμενων κανόνων. Αυτό έχει ξεκινήσει ήδη από το 2013. Επίσης, ε, στο πλαίσιο της Eurojust γίνεται συζήτηση σε επίπεδο εισαγγελέων και σύντομα θα γίνει ένας απολογισμός και εξελόγηση των πρόσφατων ευρημάτων. Τέλος, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η κατάσταση στη Λιβύη παραμένει δραματική και αυτή επηρεάζει άμεσα τις ε, επιχειρήσεις ε, έρευνας και διάσωσης στη Μεσόγειο αλλά και τις μεταναστευτικές ροές. Έχουν ε, ενταθεί εχθροπραξίες από τον Απρίλιο και μετά τις αεροπορικές επιδρομές η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος και αντιπρόεδρος Επιτροπής μαζί με τον Επίτροπο Αβραμόπουλο και τους Υπουργούς Εξωτερικών έκαναν έκκληση για άμεση δράση και εκένωση των ε, ανθρώπων από ε, αυτά τα μέρη που επλήγησαν στην Λιβύη. Χρειάζεται όμως και συνεργασία με τις αρχές τη Λιβύη. Οι ενέργειές μας στη Λιβύη συνεχίζουν να γίνονται μέσω του πλαισίου ε, συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωση και Λιβύης και της σχετικής ε, Task Force. Έτσι προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μία δομή συγκέντρωση και αναχώρησης μεταναστών στην Τρίπολη όπου θα παρέχεται προστασία. Μέσω αυτής της δομής θα ξεκινάει η διαδικασία μεταγκατάστασης και ε, υπάρχει μια, εθελο, μια προσπάθεια εθελοντική επανεγκατάσταση 55.000 μεταναστών οι οποίοι θα λάβουν την απαραίτητη στήριξη εφόσον επιλέξουν να επιστρέψουν. Επίσης, ε, στόχος είναι να μειωθούν οι επικίνδυνες και διελεύσεις ε, από τη θάλασσα, οι οποίες οδηγούν σε απώλεια ανθρώπινων ζώων λόγω της ε, πεποίθησης που υπάρχει ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Χρειάζεται λοιπόν να εντείνουμε τις προσπάθειές μας, χρειάζεται να δώσουμε αξιόπιστες εναλλακτικέ λύσεις, αλλά αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας. Χρειάζεται μια συνεργασία ε, όλων των ε, χωρών προέλευσης, χωρών διέλευσης και ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Χρειάζεται μια ολοκληρωμένη στρατηγική αντιμετώπιση της μετανάστευσης από αντιμετώπιση των αιτίων, από καταπολέμηση της ε, παράνομης διακίνησης ε, και αυτά λοιπόν. Από μένα σε ευχαριστώ πολύ. And, uh... Ήταν πολύ σαφής οι δηλώσεις σας και πραγματικά σεβαστήκατε το χρόνο, οπότε μπορούμε να περάσουμε και στο Τόμας Μόλνερ που είναι εκπρόσωπος υπηρεσίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα που θα μας δώσει κάποια στοιχεία για την ανθρώπινη διάσταση τραγωδίας αυτή στην Μεσόγειο. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε το λόγο. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή που βρίσκομαι κοντά σας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Να σας πω αξιότιμοι προσκεκλημένοι κυρίες και κύριοι, όπως είδατε στην οθόνη σας, θα μιλήσω για τις νομικές πτυχές υποχρέωσης έρευνα και διάσωσης, όπως περιγράφονται από το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο. Μιλάμε λοιπόν για θέματα τα οποία είναι επιτακτικά και υποχρεωτικά από την πτυχή των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Στο θαλάσσιο πλαίσιο, ο σεβασμός του δικαιώματος στη ζωή είναι μια νομική υποχρέωση εδώ και πάρα πολύ ε, χρόνο έχουμε την υποχρέωση παροχής βοήθειας σε ανθρώπους οι οποίοι κινδυνεύουν στη θάλασσα. Δηλαδή η διάσωση στη θάλασσα δεν είναι μόνο ένα είδος ανθρωπιστικής βοήθειας, είναι κάτι παραπάνω. Είναι ξεκάθαρα μια κομβική νομική υποχρέωση η οποία ξεκάθαρα περιγράφεται στο εθνικό διεθνές δίκαιο. Το διεθνές δίκαιο, ε, θαλάσσιο διεθνές δίκαιο, υποχρεώνει τα κράτη να λαμβάνουν προληπτική ε, δράση, δράση απόκρισης και δράση έγκαιρη προειδοποίηση έτσι ώστε να αποφεύγονται οι θάνατοι στη θάλασσα και αυτό συμπεριλαμβάνει την έρευνα και τη διάσωση. Χαρτογραφώντας το νομικό ε, τοπίο διαπιστώνουμε πως έχουμε ένα σφριγιλό και σφαιρικό ε, νομικό πλαίσιο, διεθνές νομικό πλαίσιο και στον πίνακα που έχετε στην οθόνη βλέπετε τις βασικές διατάξεις υπό τις τρέχουσες διεθνείς συνθήκες. Καταρχήν, έχουμε καταρχήν τη σύμβαση κλος για το δίκαιο της θάλασσας που περιγράφει τις ξεκάθαρες, ε, τα ξεκάθαρα καθήκοντα κάθε καπετάνιου, είτε είναι ιδιωτικό είτε είναι κρατικό το πλοίο, να διασώζει άτομα τα οποία κινδυνεύουν στη θάλασσα. Αυτό έχει να κάνει λοιπόν για τα καθήκοντα του καπετάνιου. Αλλά υπάρχουν και υποχρέωσεις, υποχρέωσεις για τις κυβερνήσεις που είναι υποχρεωμένες να έχουν υπηρεσίες ε, έρευνας και διάσωσης που θα είναι αποτελεσματικές. Η UNCLOS δεν είναι μόνο δεσμευτική για όλα τα κράτη-μέλη, αλλά αυτό εντάσσεται και στην Ευρωπαϊκή Ένωμη Τάξη, μια και εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε υποκείμενοι στο διεθνής ε, δίκαιο και είμαστε συμβαλόμενο μέρος στη σύμβαση UNCLOS. Είναι κομμάτι λοιπόν της δικής μας ευρωπαϊκής νομικής τάξης. Έχουμε και άλλες διεθνείς συμβάσεις που ε, περιγράφουν πιο λεπτομερώς αυτές τις υποχρεώσεις έρευνας και διάσωσης. Σύμβαση για την ασφάλεια της ζωής στη θάλασσα, για παράδειγμα, που περιγράφει την υποχρέωση πρακτικών και ε, αποτελεσματικών υπηρεσιών διάσωσης από τα κράτη που την έχουν υπογράψει. Όλοι εμείς είμαστε συμβαλόμενα μέρη. Επίσης, έχουμε τη Διεθνή Σύμβαση που είναι συγκεκριμένη για τη θαλάσσια έρευνα και διάσωση, που εισάγει ένα ε, συνολικό ε, καθεστώς για το συντονισμό της διάσωσης, αλλά και περιγράφει τις υποχρεώσεις των κρατών, έτσι ώστε να έχει το καθένα ξεχωριστά ε, περιοχές για τις οποίες αναλαμβάνει την υποχρέωση διάσωσης και έρευνας και έχουμε και παραπάνω λεπτομέρειες που περιγράφονται και πάνε πιο μακριά από τι αρχικέ διατάξει, όπου λέμε η συνδρομή που πρέπει να παρέχει σε οποιονδήποτε κινδυνεύει στην α, ε, ε, θάλασσα δεν επηρεάζεται ούτε από τι ε, περιστάσει από τι οποίε βρίσκεται το πρόσωπο, ούτε από την υπηκότητα, ούτε από το που. Έχουμε επίση και τη διάσωση τη Σύμβαση για τη Διάσωση που περιγράφει τις ίδιες υποχρεώσεις ε, λεπτομερώς, αλλά αυτή δεν έχει κυρωθεί τόσο εκτεταμένα. Τι λέει λοιπόν το ευρωπαϊκό δίκαιο σχετικά. Έχουμε μπροστά μας τον κανονισμό για τα θαλάσσια σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ε, εφαρμοστέος άμεσα, είναι ε, δευτεροβάθμιο νομικό εργαλείο και αυτό ε, υποχρεώνει τα κράτη-μέλη στην περίπτωση που συνεργάζονται με τη Frontex στη θάλασσα. Είναι παρόλα αυτά περιορισμένο αλλά συγκεκριμένο, γιατί έχουμε παραπάνω τις διεθνείς υποχρεώσεις, τις συμβάσεις, τις συνθήκες και έχουμε παράλληλα και αυτό το βασικό ζήτημα που είναι η συνδρομή χωρίς καθυστερήσεις οποιοδήποτε κινενεύει στη θάλασσα. Είναι σημαντικό να δούμε το εκτιμώντα 14 τούτου του κανονισμού που περιγράφει πως ο καπετάνιος δεν θα πρέπει να διώκεται ποινικά για οποιαδήποτε διάσωση ανθρώπου που κινδυνεύει στη θάλασσα και που έχει ε, μεταφερθεί σε ασφαλές καταφύγιο. Επίσης, τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα καλύπτουν αυτές οι υποχρεώσεις, βρίσκονται στο εκτιμώντας 15 και τονίζουν πως τα άτομα τα οποία σώζονται θα πρέπει να παραδίδονται σε ασφαλή τόπο. Και αυτό αποτελεί ουσιαστικό σημείο όλων των παραπάνω. Περνάμε λοιπόν και στα επιχειρησιακά του κανονισμού. Εδώ έχουμε μία φωτογραφία, άρθρο 9. Συζητάμε λεπτομέρειες το πώς γίνεται η έρευνα και η διάσωση με συγκεκριμένους κανόνες και υποχρεώσεις για την παροχή βοήθειας σε όποιον κινδυνεύει στη θάλασσα και επίσης περιγράφει ε, το πώς γίνεται η κοινοποίηση της πληροφορίας στα κέντρα διάσωσης και περιγράφει τι σημαίνει το κινδυνεύει, distress στα αγγλικά. Το άρθρο 10 μιλά για την αποβίβαση και περιγράφει την έννοια ε, του ασφαλούς τόπου, place of safety, εκεί όπου καταλήγουν οι υπηρεσίες διάσωσης. Και όλα αυτά θα πρέπει να τα διαβάζει κανείς σε συνδυασμό με, τα, με την ρήτρα ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων του ο κανονισμού που μιλάει για ε, δικλείδες ασφαλείας για την αποβίβαση σε τρίτη χώρα, δηλαδή αξιολόγηση της γενικής κατάστασης στην τρίτη χώρα πριν προχωρήσει κανείς σε αποβίβαση, όπως επίσης και τα κριτήρια της αποβίβασης μαζί με άλλα σημαντικά θέματα όπως η μετεπιβίβαση ή η μεταφορά προσωπικών δεδομένων των διασωζόμενων προς μια τρίτη χώρα. Μετά έχουμε μια γρήγορη επισκόπηση των βασικών θεμάτων. Γιατί πρέπει να έχουμε μια κοινή ε, κατανόηση του τι σημαίνουν ε, νομικά μιλώντας. Το distress κινδυνεύει. Ακολουθήσουμε λοιπόν τη λογική σειρά Είμαστε λοιπόν στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μια κατάσταση όπου υπάρχει ε, λελογισμένη βεβαιότητα ότι άνθρωπος ή σκάφος κινδυνεύει με άμεσο και σοβαρό κίνδυνο και απαιτείται άμεση ε, συνδρομή. Τι είναι διάσωση παρακάτω. Ορίζεται ε, νομικά στην ίδια σύμβαση και εδώ συμπεριλαμβάνει την εξής διάταξη. Θα πρέπει να καλύπτουν οι ιατρικές των διασωζομένων και να παραδοθούν σε τόπο ασφαλείας, σε τόπο ασφαλή. Τι είναι αυτός λοιπόν ο ασφαλής τόπος, γιατί εδώ έχουμε το πυρήνα του προβλήματος. Αυτό στην σύμβαση για τη διάσωση ε, δεν περιγράφεται, αλλά περιγράφεται στις κατευθυντήριες γραμμές που έχει εγκρίνει ο IMO μέσω της Σχετικής Επιτροπής για την Ασφάλεια και Διάσωση και έχουμε μια νομικά δεσμαυτική διατύπωση στον κανονισμό για τα θαλάσσια σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέει τόπος ασφαλής είναι ένας τόπος όπου η ασφάλεια ζωή του διασωζόμενου δεν κινδυνεύει, όπου καλύπτει βασικέ ανθρώπινε ανάγκε και από την οποία μπορούν να γίνουν κάποιε διευκολύνσει διευκολύνσεις στον τελικό προορισμό, λαμβάνοντας υπόψη τον, τα θεμελιώδη δικαιώματα και σε πλήρη σεβασμό ε, των προαναφερθέντων και του διεθνούς δικαίου. Εδώ έχουμε λοιπόν την περιοχή έρευνας και διάσωσης που θα πρέπει να ορίσει κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά και να παρακολουθεί και τα κέντρα συντονισμού που είναι οι εθνικές αρχές οι οποίες είναι υπεύθυνε για το συντονισμό αυτών των επιχειρήσεων. Όλα αυτά ορίζονται μέσω δεσμευτικών διεθνών διατάξεων στο διεθνές δίκαιο και στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Τέλος, βλέπετε στην οθόνη σας ένα χάρτη. Εδώ βλέπετε τις περιοχές που έχουν οριστεί στη Μεσόγειο ε, έτσι, να έχετε μια οπτική άποψη για το τι όψη έχουν. Και θέλω να πάω στην τελευταία διαφάνεια της παρουσίασής μου, που δεν είναι όμως και λιγότερο σημαντική. Δεν θα πρέπει να αφήνουμε στην άκρη τη διάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι υποχρεώσεις υπάρχουν για να προστατεύουν τι? Να προστατεύουν τα θεμελιώδη δικαιώματα στη ζωή. Αυτό αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή Χάρτα, το δικαίωμα στη ζωή, στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, το δικαίωμα στη ζωή. Είναι ένα από τα κομβικά ε, ανθρώπινα δικαιώματα που προστατεύεται σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο. Και δεν υπονοεί μόνο πως υπάρχει η παθητική υποχρέωση να μην σκοτώνει ένα κράτος μέλος. Όχι, είναι και ενεργητική η υποχρέωση και από το 1992 η, Επιτροπή αυτής της ε, ε, Σύμβασης του ΟΗΕ τόνισε πως η προστασία του δικαιώματο στη ζωή είναι να λαμβάνονται και κάποια ενεργά μέτρα έτσι ώστε όταν απειλείται η ζωή κανείς να παρεμβαίνει. αυτό ε, προστατεύεται και από την νομολογία. Όταν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τη ζωή. Οπότε, διάσωση και έρευνα είναι τέτοιου είδου μέτρο και δεν θα πρέπει να το θεωρείτε ως κάτι διαφορετικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, υπομονή σας. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μόλμερ, τον εκπρόσωπο του Οργανισμού ε, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και ευχαριστώ που τηρήσετε και το δεκάλεπτο. Να περάσουμε τώρα στην τρίτη προσκεκλημένη μας. Έχουμε την τιμή να δώσουμε το λόγο στην Καρόρα Ρακέτε, την πλήρχο του Sea-Watch, που θα μας πει την εμπειρία της ε, στη διάσωση ζώων ε, στις Ιταλικές ακτές ε, και γνωρίζουμε όλοι πόσο προβληματικά είναι τα πράγματα εκεί. Έχετε το λόγο για 10 λεπτά κύριε Ρακέτε. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση ε, να έρθω εδώ σήμερα και την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω στην Αρμόδια Επιτροπή για την κατάσταση στην Κεντρική Μεσόγειο. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα και λυπάμαι που κάνω την ομιλία μου σήμερα στην επέτειο της έκτης επαιτίου αυτού του περιβόητου πλέον ναυαγίου στο οποίο χάθηκαν πάνω από 360 ψυχές ε, μπροστά στη Λαμπεντούσα ε, ως αποτέλεσμα μιας ε, αποστολής διάσωσης. Έχουν περάσει έξι χρόνια και αντί να προσπαθούμε να αποφύγουμε παρόμοιες τραγωδίες, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκίνησαν μια πολιτική εξωτερήκευσης των ευθυνών τους ε, και επαναπροώθησης και δίνοντας την αρμοδιότητα σε μια χώρα η οποία βρίσκεται σε πόλεμο, στη Λιβύη, παραβιάζοντας έτσι το διεθνές δίκαιο και παρόλα αυτά ε, υπάρχουν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Κοινωνίας των Πολιτών στη θάλασσα και ε, πρέπει να προσπαθήσουν να τηρήσουν την αλληλεγγύη και το σεβασμό του δικαιώματος ε, στη ζωή του καθενός που είναι θεμελιώδες δικαίωμα. Εγώ είμαι ανεξάρτητη εθελοντή που ξεκίνησε το 2016 και αποφάσισα να προσφέρω την εμπειρία μου ω πλοίαρχο. Στην πρώτη αποστολή διασώσαμε εκατοντάδε ζωέ και ε, ε, είχαμε παρέμβαση σε ένα φρικτό ναυάγιο στο οποίο συμμετείχαν και σκάφη του λιμενικού. Από ό,τι θυμάμαι το σκάφος μας ε, το είχαν περικυκλώσει πτώματα τα οποία επέπλεαν. Κάποιοι άνθρωποι είχαν πεθάνει αγκαλιασμένοι και κάποια πτώματα ήταν αχώριστα. Ο Μάικολ, ένας από τους εθελοντές μας, πατέρας τριών παιδιών, διέσωσε το σώμα ενός ε, βρέφους. Δεν μπορούσε να δεχτεί ότι δεν υπήρχε ε, καθόλου ζωή σε αυτό το μικρό πλασματάκι. Του τραγουδούσε και το αγκάλιαζε σαν να ήταν ζωντανό. Μείναμε μέχρι την αυγή, συλλέγαμε πτώματα με το πολεμικό ε, σκάφος, ε, ένα ιταλικό σκάφος, τον Ave Vega και πραγματικά ε, προσπαθούσαμε να βρούμε τα πτώματα, τα δέναμε σε ένα χέρι, σε ένα πόδι μέχρι να μπορέσουν να τα πάρουν οι διασώστες. Ε, συμμετείχα επίσης και σε ε, αποστολές παρακολούθηση του Sea Watch και πολλές φορές είδα ανθρώπους να του αφήνουμε στη θάλασσα ή να επιστρέφονται στη Λιβύη από τη χώρα από την οποία μόλις είχαν προσπαθήσει να ξεφύγουν. Καμία από αυτές τις εμπειρίες όμως δεν ε, μετάραξε τόσο πολύ ώστε να βρίσκομαι στο Sea-Watch ε, για 17 ημέρες και να πρέπει να εξηγήσω στους επιζώντες που είχαμε διασώσει ότι μία χώρα σε ειρήνη δεν τους ήθελε. Ότι η Ευρώπη, το λεγόμενο λίκνο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων δεν επέτρεπε να αγγίξουμε την ε, επικράτειά τους. Και πραγματικά ήταν πονίδιστο το γεγονός αυτό παρά ε, το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι, ε, τα θεσμικά όργανα και μη κυβερνητικέ οργανώσεις είχαν στρέψει τα μάτια τους σε εμάς, εγώ ήμουν μόνη μου με τους ανθρώπους που είχαμε διασώσει και πραγματικά αντιμετώπιζα ένα ε, φανταστικό πνευματικό πόλεμο και δεν υπήρχαν πραγματικά όρια σε αυτό τον πόλεμο. Η υπόθεση του Sea-Watch για άλλη μια φορά ε, έθεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση ενώπιον ε, των ευθυνών της. Ε, το γεγονός ότι τα κράτη-μέλη δεν είναι πρόθυμα να αντιμετωπίσουν ένα διαρθρωτικό φαινόμενο και να συμφωνήσουν για την ανακατανομή 53 ατόμων. Και έτσι υποχρεώθηκαν να μπω στο λιμάνι της Λαμπεντούσα μόνιμου με υποδέχτηκαν σαν να ήμουν ένα σκάφος που είχε πανόλι και όχι ένα σκάφος το οποίο είχε ευάλωτους και εξαντλημένους ανθρώπους. Βάσει του διεθνώς δικαίου, το Sea-Watch που μετέφερε 53 άτομα θεωρήθηκε ε, απειλή για την ε, δημόσια ασφάλεια. Υπήρχε προσοχή την οποία δεν ήθελα, ε, απειλές από ευρωπαϊκές χώρες και θεσμικά όργανα μετά από την είσοδό μου στο λιμάνι αλλά πού ήσασταν εσείς όταν ζητούσαμε βοήθεια από όλες τις επιχειρησιακές νομικές ε, οδούς, από κανάλια και από διπλωματικές οδούς και όταν η μόνη απάντηση που έλαβα για το αίτημα για έναν ασφαλή λιμένα ε, για αποβίβαση των ανθρώπων αυτών ήταν η Τρίπολη, σε μια χώρα σε πόλεμο όπου οι άνθρωποι ε, βίωναν συστηματικά παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Μετά από 17 ημέρες έπρεπε να μπω στο λιμάνι όχι για να προκαλέσω όπως το εξέλαβαν πολλοί, αλλά από ανάγκη για να, και από ευθύνη ενώπιον όλων αυτών των ανθρώπων που βρίσκονταν επί του σκάφους μου, αλλά και ευθύνη απέναντι στον εαυτό μου. Δεν είχα κοιμηθεί ούτε εγώ ούτε το πλήρωμα για μέρες και μετά μου κοινοποίησαν ότι ε, διεξάγεται ποινική έρευνα και τουλάχιστον όμω ε, μπορεί αυτό να οδηγούσε στο τέλος μια απίστευτη κατάστασης. Τελικά όμως ε, δεν έγινε τίποτα. Δεν θεώρησαν ότι ήταν ασφαλέ πλέον να είμαι εγώ υπεύθυνη για όλου αυτού του ανθρώπου που βρίσκονταν επί του σκάφου για πάνω από δύο ημέρες έπρεπε να έχουμε επιπλέον περιπολίες ε, στο σκάφος για να αποφύγουμε το μοιραίο, τις ε, θεωρούσαμε περιπολίες αυτοκτονίες. Άρχισε να χάνεται η εμπιστοσύνη και να απελπίζεται ο κόσμος και πραγματικά φοβόμουν ότι θα μπορούσε να συμβεί το ανεπανόρθωτο και εγώ ως πλήρχος είχα υποχρέωση να τους πάω σε κάποιο ασφαλές μέρος και μάλιστα είχα καθυστερήσει για πάρα πολλές. Ζήτησα τη στήριξη των αρχών συνεχώς επί 17 ημέρες και τέλος χρειάστηκε να το κάνω μόνη μου. Ήμουν νομικά υπεύθυνη για τη ζωή άλλων ανθρώπων ως πλήρχος, αλλά πέραν αυτού ήμουν και υπεύθυνο ως άνθρωπος για τη ζωή τους. Η κατάσταση θα μπορούσε να είχε επιληθεί πολύ νωρίτερα την ημέρα μετά από τη διάσωση υπήρχε ένας δήμος ε, από ένα δίκτυο 60 πόλεων αλληλεγγύης είχαν προσφερθεί να, δεχ, να υποδεχτούν τους ανθρώπους που είχαμε διασώσει. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει δυνατότητα να υποδεχθούμε αυτούς τους ανθρώπους. Η δική μας περίπτωση, όπως και η περίπτωση άλλων μη κυβερνητικών οργανώσεων, ε, ζητά ε, ευθύνη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να γίνονται αυτά βάσει νόμου και δεν μπορούμε να είμαστε υπό όρου σε ad hoc διαπραγματεύσεις ε, ανάλογα με τη βούληση του κάθε κράτους μέλους και κάθε φορά ε, μπορεί να άγεται και να φέρεται από συγκεκριμένα συμφέροντα. Αυτό δεν είναι ούτε βιώσιμο αλλά ούτε και αξιόπιστο. Χρειάζεται μία αλλαγή του συστήματος. Ε, μία προσωρινή συμφωνία επανεγκατάστασης ουσιαστικά θέλει απλώς να επιστρέψει οι ανθρώπους και όχι να τους υποδεχθεί. Ε, και δεν υπάρχουν κριτήρια για την επανεγκατάσταση. Ε, λαμβάνουν υπόψη μόνο ε, ανθρώπους οι οποίοι διασώζονται από μη κυβερνητικέ οργανώσεις, δεν λαμβάνονται υπόψη εμπορικά σκάφη και τη βούληση κάποιων δήμων να τους υποδεχθούν. Πρέπει να ε, προφυλάξουμε το δικαίωμα των ανθρώπων να ζητούν άσυλο και να υπάρχουν συγκεκριμένοι λιμένες αποβίβασες και να υπάρχουν και ανθρωπιστικοί διάδρομοι από τη Λιβύη. Χρειάζεται μεταρρύθμιση του κανονισμού του Διβλίνου, η οποία έχει καθυστερήσει πάρα πολύ και θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό στι επόμενε εβδομάδε. Ο καλύτερο τρόπο όμω για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει πρόσβαση σε διαδικασίε ασύλου σημαίνει ότι θα πρέπει να φτάνουν με ασφάλεια και με νόμιμο τρόπο στην Ευρώπη. Δεν χρειάζεται μόνο μεταρρύθμιση του κανονισμού του Διβλίνου, χρειάζεται και μια ασφαλής οδός. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εγώ ακόμα είμαι υποέρευνα. Ε, υπάρχουν δύο ποινικέ διαδικασίες ε, εναντίον μου στην Ιταλία για τη διέσωση ανθρώπου ε, στη θάλασσα. Εγώ δεν ανησυχώ γιατί οι δράσεις μου ήταν βάση νόμου και ηθικές ε, και εγώ προασπίζομαι τα ανθρώπινα δικαιώμα. Η απόφαση του δικαστή για τη σύλληψή μου είναι ότι ήταν το καθήκον μου. Το πρόβλημα είναι ότι το Sea-Watch 3 έχει αλλάξει και έχει γίνει μια διοικητική κατάσχεση. Ε, πρόσφατα ε, απελευθερώθηκε από το δικαστήριο του Αγκριτζέντο, αλλά ε, λόγω ε, νόμου για την ασφάλεια δεν μπορεί να βρίσκεται στη θάλασσα ακόμα. δεν μπορεί να δίνουμε την ευθύνη στις λιβικές αρχές, οι οποίες δεν είναι υπόλογες ενάντια σε κανέναν και δεν ξέρουμε και πόσοι άνθρωποι μένουν χωρίς ε, συνδρομή. Την περασμένη Κυριακή είχαμε την ημέρα μεταναστών ε, και προσφύγων, ενώ είχαμε αφήσει 80 ώρες ανθρώπους ε, στη μέση της θάλασσας πριν τους επιστρέψουμε στη Λιβύη, όπου πραγματικά υποφέρουν. Ενημερώθηκαν οι αρχές, αλλά και αυτή η περίπτωση θα προστατεύεται και πάλι από τη μορισία. Κάθε φορά που ένα σκάφος μιας κυβερνητική οργάνωση ε, κάνει το καθήκον του και διασώζει οποιονδήποτε στη θάλασσα, ξεκινούν ποινικέ διαδικασίε αν δεν είναι αυτό στρέβλωση της δικαιοσύνης, τι είναι. Τιμωρούνται πολίτες οι οποίοι υπερασπίζονται το κράτος δικαίου και προστατεύουν ε, μια παράνομη κρατική πρακτική. Η κεντρική θάλασσα της Μεσογείου γίνεται ένα έρημο νεκροταφείο και ε, άνθρωποι οι οποίοι ε, επιστρέφονται και υποχρεώνονται να πάνε σε μια ασφαλά μέρη και η διάσωση ποινικοποιείται.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 Thank Σας ευχαριστούμε κυρία Ρακέτε. Το χειροκρότημα που δεχτήκατε νομίζω πως είναι ένα δείγμα της εκτίμησης που έχουμε στο έργο σας. Έχετε δείξει τη μεγάλη προσωπική σας δέσμευση. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ. Ε, σίγουρα θα ακολουθήσει και γύρω ερωτήσεων ε, προς εσάς μόλις ολοκληρώσουμε τις παρεμβάσεις των προσκεκλημένων μας. Σε αυτή την ακρόαση λοιπόν για την έρευνα και διάσωση. Θα συνεχίσουμε τώρα με τον τέταρτο προσκεκλημένο, τον ε, Αντρέα Τασάρα από την Ιταλική Ακτοφυλακή, ο οποίος συμμετέχει ενεργά σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να ακούσουμε και τη δική σας μαρτυρία και σας ε, καλωσορίζουμε στην Επιτροπή μας. Έχετε το λόγο για 10 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα συνεχίσω στα Ιταλικά, κυρίε και κύριοι. Κύριε Πρόεδρε, εξότιμα μέλη τη Επιτροπής, ε, θα ήθελα να απευθύνω χαιρετισμό και εξ ονόματος του Ναβάρχου Γενικού Διευθυντή της Ακτοφυλακής ε, και α, εκ μέρους των 11.000 ανδρών και γυναικών ε, μελών της ακτοφυλακής της Ιταλίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση εδώ, για να συμβάλλουμε και εμείς από τεχνική σκοπιάς ε, και να σας παρουσιάσουμε την οπτική ε, της Ιταλικής ακτοφυλακής ε, για να κατανοήσουμε λίγο καλύτερα το φαινόμενο της διάσωσης στη θάλασσα, στην κεντρική Μεσόγειο. Η Από το 1998 μέχρι σήμερα η Ιταλική ακτοφυλακή έχει διασώσει περίπου ένα εκατομμύριο ανθρώπους. Ο προλαλής αναφέρθηκε σε όλες τις συμβάσεις ε, και ε, τις ε, νομοθεσίες που διέπουν τη διάθεση στη θάλασσα και κυρίως μας ενδιαφέρει η σύμβαση του Αμβούργου που καθορίζει υποχρεώσεις και για τους κυβερνήτες του ναυτικού αλλά και για τις δυνάμεις διάσωσης και μάλιστα η διάσκεψη ΣΑΡ ε, προβλέπει ότι θα πρέπει να δίνεται βοήθεια σε κάθε άτομο που βρίσκεται σε κίνδυνο στη θάλασσα χωρίς διάκριση εθνικότητας, ε, το καθεστώς αυτού του ανθρώπου ή τις συνθήκες ε, μέσω των οποίων βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος στη θάλασσα. Επίσης, η Σύμβαση ΣΑΡ προσπαθεί να προωθήσει και τη συνεργασία μεταξύ κρατών, την προωθεί μάλιστα για να τηρηθεί η αρχή της ακαιρεότητας ε, των υπηρεσιών και ζητά όλα τα, από όλα τα κράτη να έχει μια περιοχή ευθύνη στην οποία θα πρέπει να είναι αρμόδια για τη διάσωση. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν κυρώσει όλες οι χώρες τη σύμβαση αυτή και οι κατευθυντήριες γραμμές ε, του IMO προβλέπουν ότι το πρώτο κέντρο ε, διάσωσης το οποίο λαμβάνει είδηση για πιθανή επίγουσα κατάσταση είναι υπεύθυνο για να λάβει τα πρώτα μέτρα ε, διάσωσης για την κατάσταση και ακόμα και αν βρίσκεται εκτός από την περιοχή της δικής του ευθύνης. Αυτό μέχρι του σημείο που το κέντρο διάσωσης που είναι αρμόδιο ανα, την, ε, να αναλάβει την ευθύνη για την ε, περίπτωση αυτή. Και αυτό καθορίζει λοιπόν ότι όποιος ε, βρίσκεται ε, επί στη θάλασσα θα πρέπει να κοινοποιεί στις αρμόδιες αρχές η διάσωση των ανθρώπων δεν σημαίνει ότι ολοκληρώνεται η επιχείρηση, γιατί η επιχείρηση μπορεί να θεωρηθεί ότι ολοκληρώθηκε αποκλειστικά μόνο με την αποβίβαση αυτών των ανθρώπων σε έναν ασφαλή χώρο, το λεγόμενο place of safety. Ε, γι' αυτό ακριβώς ε, ο χώρος και η υποχρέωση να βρεθεί αυτός ο χώρος ασφαλείας ε, σε συνεργασία με όλες τις πιθανόν ενδιαφερόμενες αρχές εμπίπτει στο κέντρο το οποίο ανέλαβε την ευθύνη του συντονισμού. Τώρα, οι εγκληματικές οργανώσεις οι οποίες διακινούν ανθρώπους εκμεταλλεύονται προς όφελός τους τέτοιες ε, διατάξεις, ε, υποχρεώνοντας ε, και κάποιες φορές δια της βίας κάποιους ανθρώπους να βρεθούν στα σκάφους τους, δημιουργώντας ε, προβλήματα ε, κινδύνου, distress όπως είπαμε προηγουμένως ε, και φυσικά υποχρεώνονται κάποιοι να διασώσουν αυτούς τους ανθρώπους. Αυτές οι διαδικασίες αποδεικνύουν ότι η σύμβαση ΣΑΡ όπως και άλλες υποχρεώνουν να διασώζουμε για κάποιες τυχαίες ε, ε περιπτώσεις ε, και όχι γιατί κάποιος δημιουργεί συνθήκες κινδύνου στη θάλασσα. Η μόνη χώρα που παρά το γεγονός ότι δεν έχει κυρώσει τη σύμβαση του Αμβούργου, παρόλα αυτά κύρωσε μάλλον τη σύμβαση, αλλά δεν έχει καθορίσει το χώρο ΣΑΡ ε, που τις όπου θα προσφέρει η διάσωση είναι η Τινησία. Η Λιβύη έχει κυρώσει τη Σύμβαση του Αμβούργου και έχει υποσήμως ε, διακηρύξει την περιοχή Ευθύνη τη ε, στις 14 Δεκεμβρίου του 2017. Την περιοχή αυτή μπορείτε να τη βρείτε και στο Global Integrated Shipping System που είναι το GSIS ε, του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Όσον αφορά την οργάνωση διάσωσης της Ιταλίας, ο το Υπουργείο Μεταφορών είναι το αρμόδιο. Η ακτοφυλακή είναι αρχή η οποία είναι αρμόδια για την διάσωση στη θάλασσα και η οργάνωση ε, γίνεται στα 8 χιλιόμετρα των ε, Ιταλικών ακτών και σε 500 ε, τετραγωνικά χιλιόμετρα περιοχής στη Μεσόγειο. Για το μεταναστευτικό φαινόμενο, το βασικό στοιχείο είναι ότι βρίσκονται σε κίνδυνο ε, οι μετανάστες ε, με τα σκάφη με τα οποία κυκλοφορούν. Είναι σκάφη τα οποία είναι κάκης της κατασκευής, ορισμένες φορές είναι υπερφορτωμένα, γεμάτα με γυναίκες και παιδιά, χωρίς ε, τα απαραίτητα μέσα ασφαλείας. Οι δυνατότητες διάσωσης αλλά μας ενδιαφέρει, είναι σημαντικές, αλλά μας ενδιαφέρει και ο έλεγχος των συνόρων. Η γεωγραφική περιοχή έχει και ευαίσθητες ε, κοινωνικοπολιτικές προεκτάσεις και φυσικά πρέπει η Ιταλική Ακτοφυλακή να συντονίσει ορισμένες φορές ακόμα και εκτός από τη δική της την δικαιοδοσία ε, αρκετά σκάφη τα οποία είτε είναι δημόσια είτε είναι ιδιωτικά. Ε, η κατάσταση επιδεινώνει και από το γεγονός ότι υπάρχουν και ε, αρχές ε, κυβερνητικές από αρκετές χώρες και υπάρχουν και αρκετά σκάφη τα οποία διαχειρίζονται μη κυβερνητικές οργανώσεις. Όλα αυτά τα σκάφη, αυτές οι μονάδες, ανεξάρτητα από το σκοπό δραστηριότητές τους, ε, είναι υποχρεωμένα να σέβονται το άρθρο 98 της ε, σύμβαση του Μεντέγκο Μπέι, βάσει του οποίου ο πλοίαρχο οποιοδήποτε σκάφο πρέπει να παρέχει άμεση βοήθεια σε όποιον βρίσκεται σε κίνδυνο και να συνεργάζεται με τα κέντρα ΣΑΡ. Ο ασφαλής χώρος, ε, το place of safety, καθορίζεται στη συνέχεια μετά από τη διάσωση. Υπάρχουν ε, ε, συγκεκριμένες προεκτάσεις και σε ανθρωπιστικό επίπεδο και κάποιες διεθνείς προεκτήσεις. Ε, τα όσα σας λέω ε, επαναλήφθηκαν και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που ε, υποχρεώνει και σεβασμό, σε σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και επομένως ε, δεν θα πρέπει τα κράτη να κάνουν οτιδήποτε ε, θεωρηθεί επαναπροώθηση και ταυτόχρονα να εξασφαλίσουν και την αποβίβαση αυτών των ανθρώπων αφού τους έχει δοθεί βοήθεια σε έναν ασφαλή χώρο, ένας χώρος ο οποίος ε, θα ανταποκρίνεται όχι μόνο στις βασικές πρώτες ανάγκες, αλλά θα πρέπει να γίνονται σεβαστά και τα θεμελιώδη δικαιώματά τους και να υπάρχει πρόσβαση σε μια δίκαιη και αποτελεσματική διαδικασία ασύλου. Το να βρεθεί ένας ασφαλής χώρος είναι μια πολύ περίπλοκη διαδικασία. Εμπίπτει στην αρμοδιότητα του κέντρου διάσωσης, ε, το οποίο συντονίζει τις επιχειρήσεις στη θάλασσα και περιλαμβάνει και αρκετούς άλλους φορείς. Ο σκοπός φυσικά των κανόνων που προωθήθηκαν ε, ε, το 2008 είναι να ε, συνοδεύει την υποχρέωση διάθεσης του πλοιάρχου και ε, να δίνει και οποιαδήποτε συνδρομή. Ε, οι χώρες λοιπόν στις οποίες γίνεται η πρώτη λήψη του, του σήματος για την ανάγκη για διάσωση θα πρέπει να βρούνε στη δική τους την επικράτεια ένα χώρο ασφάλειας. Επίσης, η υποχρέωση αυτή προκύπτει και από την ε, πλήρη θαλάσσια δικαιοδοσία ενός ε, παράκτιου κράτους. Η γεωγραφική θέση της Ιταλίας ε, την κάνει να είναι τελικός προορισμός των μεταναστευτικών ορών και έτσι το Υπουργείο Εσωτερικών της Ιταλίας έχει την ευθύνη να συντονίσει μέσω και των Δήμων ε, την υποδοχή επί ξηράς και να συμμετέχουν και αρκετές ε, δημόσιες αρχές. Ε, υπάρχουν επίσης πολλές διεθνείς οργανώσεις, ο IMO, η Frontex κλπ. Επίσης, πέρα από το γεγονός ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη και τι προβληματικά στοιχεία υπάρχουν κυρίως όσον αφορά την, το σκάφος, ε, θα πρέπει να υπάρχει και συντονισμός από το Κέντρο Διάσωσης και με το Υπουργείο Ιστορικών. Για να προχωρήσουμε όλες αυτές τις διαδικασίες βέβαια υπάρχουν κάποιες επιχειρησιακές διαδικασίες οι οποίες θεωρούνται ο κανόνας και πρέπει να είναι ο τρόπος με τον οποίο θα συνδιαλεγόμαστε με τα, τους αρμόδιους του Υπουργείου Εσωτερικών. αφού οι στιγμή έχουν διασωθεί οι άνθρωποι για να δούμε πού θα φτάσει ε, το σκάφος. Ε, τώρα, το τι γίνεται με τις λιβικές αρχές ε, και τη διαδικασία σταθεροποίησης της Λιβύας ε, και τη συνεργασία που αποφασίστηκε με την ε, προσωρινή κυβέρνηση της Λιβύας η οποία αναγνωρίστηκε από τα Ηνωμένα Έθνη λαμβάνει υπόψη της και τις συμφωνίες που υπάρχουν μεταξύ Ιταλίας και Λιβύης και στα πλαίσια βέβαια της ισχύουσας διαδικασίας μέσω των ψηφιμάτων ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Υπάρχουν πάρα πολλές ε, ε, αποφάσεις δικαστηρίων. Υπάρχει, για παράδειγμα, και τα όσα ε, κάνει και η ακτοφυλακή για να εκπαιδεύσει ε, της, τη λιβική ακτοφυλακή στα πλαίσια της Uniformed. Επίσης, υπάρχει και ένα κέντρο συντονισμού της Λιβύης, το οποίο προώθησε η Γενική Διεύθυνση HOME και η εξωτερική υπηρεσία δράσης ε, για να λάβει υπόψη της και κάποιες δραστηριότητες. Ε, δραστηριότητες ε, οι οποίες επέτρεψαν στη Λιβύη να καθορίσει το δικό τους χώρο ευθύνης για την έρευνα και τη διάσωση στη θάλασσα και να δημοσιεύσει τα στοιχεία που αφορά τον Εθνικό Οργανισμό στο GSIS του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Να πω ότι σήμερα η εκτοφυλακή συμμετέχει και σε νέο πρόγραμμα δημιουργία ικανοτήτων για να προσπαθήσουν να αναπτύξουν και να βοηθήσουν τη Λιβύη, που ε, τίτλο ε, υποστήριξη για την ένταξη και τη διαχείριση που ε, καθοδηγείται από το Υπουργείο Ιστορικών της Ιταλίας και φυσικά συνοδεύεται και από τη βοήθεια της Ιταλικής Ακτοφυλακής. Η Ακτοφυλακή λοιπόν ανταποκρίθηκε στην κατεπίγουσα αυτή ανάγκη και προσάρμοσε την ομοθεσία της σε μια διαδικασία άνευ προηγουμένου και από το 2013 στο 2017 ανέλαβε να κάνει διάσωση στη θάλασσα σε μια περιοχή που ουσιαστικά αντιστοιχεί στο 1 τρίτο της Μεσογείου. Λόγω όμως της κατάστασης δεν μπορεί παρά να ζητάμε μια κοινή προσέγγιση σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και να αναγνωρίσουμε ναι μεν ότι η Ιταλία έχει κάνει μια τεράστια προσπάθεια αλλά πρέπει να προχωρήσουμε γιατί αυτή η ασθένεια δεν γεννάται στη θάλασσα ε, αναπτύσσεται στην ξηρά. Επομένως πρέπει να δράσουμε εκεί. Σας ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη αν μακρηγόρησα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ σας ευχαριστώ, πλήρχε Ανδρέα Τασάρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η μαρτυρία σας είναι ευπρόσδεκτη και μπορείτε να είστε βέβαιος ότι η ακτοφυλακή και η δουλειά της αναγνωρίζετε από όλους εκείνους που έχουν μια κάποια εμπειρία επιτόπου, αναγνωρίζουμε τι έχετε κάνει για ε, το θέμα αυτό τα τελευταία χρόνια και για τη διάσωση ζών στη θάλασσα. Όπως βλέπετε και στην οθόνη σας έχουμε εδώ τον εκτελεστικό διευθυντή της Frontex. της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας δηλαδή για την προστασία των συνόρων με έδρα την Βαρσοβία. Είστε προσκεκλημένος για να μοιραστείτε μαζί μας τις απόψεις σας για το θέμα αυτό έτσι ώστε να ακολουθήσει διάλογος. Έχετε λοιπόν το λόγο για 10 λεπτά και να πω ότι ο κύριος ε, Λετζερή ως ε, εκτελεστικός διευθυντής της Frontex δεν έχει δυστυχώς πολύ χρόνο για να ανταλλάξει απόψεις μαζί μας. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω ο πρώτος γύρος των ερωτήσεων ε, να ε, απευθυνθεί στον κύριο Λεζερή. Διότι πρέπει να φύγει λοιπόν αμέσω ε, μετά. Μετά θα ακολουθήσει και δεύτερο γύρο ερωτήσεων. Γι' αυτό λοιπόν ε, σα δίνω το λόγο και σα παρακαλώ να κρατήσετε το χρονό ομιλία. Κύριε Λεζέρε, έχετε το λόγο για 10 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ εσάς και την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να ε, συμμετάσχω έστω και με αυτόν τον τρόπο στην ακρόαση αυτή. Όπως είπε και ο Πρόεδρος, αυτή την ε, ώρα γίνεται μία έκτακτη συνάντηση στην ε, Βαρσοβία, στη Frontex, αλλά ήθελα να είμαι παρόν και να συμμετάσχω στην ε, ακρόαση. Γι' αυτό λοιπόν βρίσκομαι εδώ. Οι συζητήσεις που διεξάγονται σήμερα το πρωί στην ε, Βαρσοβία νομίζω πως ε, θα πρέπει να δώσουν την δυνατότητα να εξερευνήσουμε τις δυνατότητες που έχουμε στο εφιστάμενο νομικό πλαίσιο ε, σε ό,τι αφορά τους πόρους της ε, Frontex. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ε, μόνιμο σώμα ακτοφυλακής, που είναι το πιο σημαντικό τμήμα του σχετικού κανονισμού, αποτελεί το πιο σημαντικό κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακή. Ο ρόλος μας είναι να ε, παρέχουμε συνδρομή στα κρατημέλη στις ε, δικές τους επιχειρήσεις έρευνα και διάσωση. Όπως γνωρίζετε, ή μπορεί και να μην το γνωρίζετε, η Frontex έχει αναγνωριστεί από τον ε, Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό το 2018 ως σημαντικός παράγοντας. Έχουμε διασώσει πάνω από 88.000 ανθρώπους στη θάλασσα. Αυτός είναι ο συνολικός ε, αριθμός των διασωθέντων. Και από τον Ιανουάριο μέχρι τον Οκτώβριο του 2018 διασώσαμε 60.000 ανθρώπους. Φέτος, μέχρι τώρα, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων μας, έχουμε διασώσει πάνω από 30.000 ανθρώπους στη θάλασσα. Και αυτό έγινε σε πάνω από 1.100 επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις μας έχουμε διασώσει χιλιάδες ανθρώπους, πάνω από 20.000 διασωθέντες στην επιχείρηση Ποσειδών στην Ελλάδα. Φέτος έχουμε διασώσει σχεδόν 15.000 ανθρώπους στην Ισπανία και σχεδόν 2.000 ανθρώπους ε, στο πλαίσιο της επιχείρησης Θέμης στην Κεντρική Μεσόγειο. Όπως γνωρίζετε, η Frontex συμμετέχει επίσης ε, στο δίκτυο Ευρωπαϊκών ε, Οργανισμών Ναυτιλίας και με τις οποίες μοιράζεται μια κοινή εντολή διαφύλαξη των θαλάσσιων συνόρων. Γίνονται εργαστήρια, γίνονται ασκήσεις, ειδικές ε, δραστηριότητες και εκπαιδευτικά σεμινάρια, τα οποία αποτελούν κεντρικό κομμάτι αυτής της ευρωπαϊκής συνεργασίας με τους άλλους ε, οργανισμούς και με τις ε, εθνικές ακτοφυλακές. Η Frontex σιγά σιγά στρώνει το δρόμο για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής Ταυτότητα που χαρακτηρίζει την ε, ακτοφυλακή και τι επιχειρήσει έρευνα και διάσωση και θα παραμείνει κεντρικό κομμάτι των καθηκόντων μας. Το νομικό πλαίσιο της ε, Frontex περιέχει συγκεκριμένους κανόνες για την ε, παρακολούθηση στη θάλασσα και τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης καθώς και τους κανόνες αποβίβασης. Υπάρχουν επιχειρησιακά σχέδια για κάθε μία επιχείρηση μας. Ε, είναι σχέδια πάνω στα οποία έχουμε συμφωνήσει με το κράτος ε, μέλος που φιλοξενεί τις ε, επιχειρήσεις αυτές. Γι' αυτό λοιπόν εμείς έχουμε τα νομικά όπλα για να διεξάγουμε αυτές τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Θα ήθελα όμως να σας υπενθυμίσω ότι η Frontex δεν μπορεί να προτείνει η ίδια τη διεξαγωγή μιας επιχείρησης και δεν μπορεί να διατάξει την ανάπτυξη θαλάσσεων ε, δυνάμεων και σκαφών χωρίς πρώτερη έγκριση για αποβίβαση. Έτσι λοιπόν αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να στείλουμε σκάφη, δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε μια επιχείρηση εάν δεν υπάρχει πρώτερη έγκριση για το σημείο αποβίβασης, ε, πιθανώς ε, παράνομων μεταναστών που διασώζονται στη θάλασσα. Βέβαια, δεν υπάρχει νομικό κενό εδώ. Το δίκαιο της θάλασσας είναι σαφέστατο και ο διασωθέντας πρέπει να μεταβεί στο ε, πιο κοντινό ασφαλές ε, λιμάνι. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να γίνει μια διευκρίνηση. Η Frontex ως ε, Οργανισμός ε, Συνόρων και ε, Ακτοφυλακής δεν είναι μια υπηρεσία που αναλαμβάνει μόνο επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Υπάρχουν ε, άλλες σχετικές υπηρεσίες. Η Frontex δεν κάνει λοιπόν μόνο αυτό, έχει και άλλες πολύ σημαντικές ε, λειτουργίες και καθήκοντα συνοδεύει ε, τις αρχές επιβολής του νόμου και εφαρμόζει το δίκαιο της θάλασσας, ε, διεξάγονται επιχειρήσεις κατάσχεση κατάσχεσης ε, ναρκωτικών, ε, κατα, πολέμησης παράνομης διακίνησης όπλων και άλλων εγκληματικών δραστηριοτήτων. Πολλές φορές προκύπτει ένα ερώτημα το οποίο θα ήθελα να απαντήσω. Ακούγεται λοιπόν ότι η Frontex έχει εντολή να συντονίσει κοινέ επιχειρήσεις οι οποίες θα έχουν αποκλειστικό ε, σκοπό την έρευνα και τη διάσωση. Ο λόγος γι' αυτό είναι επειδή δεν υπάρχει ευρωπαϊκή αρμοδιότητα για την έρευνα και διάσωση. Νομικά αυτό είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Αυτό που στην πράξη συμβαίνει είναι διάφορες επιχειρήσεις παρακολούθησης ε, των συνόρων και στο πλαίσιο αυτών των επιχειρήσεων έχουμε τη δυνατότητα να στηρίξουμε ε, και άλλες επιχειρήσεις και να αναλάβουμε συντονιστικό ρόλο. Γι' αυτό τον λόγο καταφέραμε να διασώσουμε ε, με επιτυχία πάνω από 38.000 ανθρώπους φέτος μόνο. Να σας εξηγήσω λίγο πώς λειτουργεί αυτό επιχειρησιακά. Η ανάπτυξη λοιπόν μία επιχείρησης έχει μια εντολή που αφορά την παρακολούθηση των συνόρων. Υπάρχει μια ιεραρχία. Εμείς πάντα εκτελούμε εντολές ε, υπό τις εθνικές αρχές του κράτους μέλους που μας φιλοξενεί. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Κάθε κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, έχει μία εθνική αρχή που συντονίζει τις δράσεις έρευνας και διάσωσης και μία περιφερειακή αρχή που διεξάγει ε, παρακολούθηση στα σύνορα. Οι δραστηριότητες λοιπόν αυτές που αφορούν μόνο την παρακολούθηση των σύνορων ε, στις οποίες συμμετέχουμε ε, είναι δραστηριότητες ε, όπου εμείς παίζουμε δευτερεύοντα ρόλο. Ενεργούμε υπό τις εντολές ε, της Εθνικής Αρχής. Μετά, από εμά η ιεραρχία αλλάζει και σε περιπτώσει έρευνα και διάσωση, υπεύθυνο είναι το κέντρο έρευνα και διάσωση στη θάλασσα. Όταν δεν ολοκληρώνεται μια, μια επιχείρηση έρευνα και διάσωση, εμεί ε, συνεργαζόμαστε με το κέντρο συντονισμού του κράτου ε, μέλου που μα φιλοξενεί. Αυτό γίνεται σύμφωνα πάντα με το δίκαιο τη θάλασσα. Οφείλουμε όμως να πούμε ότι η έρευνα και η διάσωση θα πρέπει να παραμείνουν εξαίρεση και να μην γίνουν κανόνας στις ε, δραστηριότητές μας. Αυτό πολύ συχνά ε, είναι αυτό που συμβαίνει στην κεντρική Μεσόγειο. Δεν πρέπει ούτε να δεχτούμε ούτε να ανεχόμαστε ε, διακινητές και λαθρεμπόρους οι οποίοι κάνουν κατάχρηση των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης για να κάνουν τις ε, δουλειές τους και να αποκομίζουν τεράστια κέρδη παίζοντας με ανθρώπινες ζωές αυτών των μεταναστών. Θεωρούμε πως έχουμε ανθρωπιστικό καθήκον να αντισταθούμε σε αυτό που συμβαίνει. Όμως έχουμε και ένα άλλο καθήκον ε, ως, και εγώ προσωπικά ως επικεφαλής ε, της ε, υπηρεσίας αυτής να πω ότι οφείλουμε να συνεχίσουμε τον αγώνα κατά του διασυνοριακού εγκλήματος και να προσπαθήσουμε να εξαρθρώσουμε τα εγκληματικά δίκτυα. Οφείλουμε να πούμε ότι ζούμε ε, καταστάσεις στην κεντρική Μεσόγειο, οι οποίες πολλές φορές είναι τεχνητά δημιουργημένες από αυτά τα ε, εγκληματικά δίκτυα. Και πώς από τη στιγμή που ο μετανάστης πέφτει στα χέρια λαθρεμπόρων και διακινητών, ε, αναπόφευκτα θα γίνει αντικείμενο έρευνας και διάσωσης. Και αυτό συνεπάγεται όλους τους κινδύνους που φαντάζεστε. Αυτή λοιπόν είναι η οπτική γωνία της ε, Frontex. Υπάρχει ένα έντονο στοιχείο έρευνας και διάσωσης ε, στις δραστηριότητές μας και νομίζω πως είναι σαφές ότι η Frontex ε, στο πλαίσιο των καθηκόντων της έχει αφιερώσει κονδύλια στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Όπως σας είπα και πριν, οι οποίε υπάγονται στο γενικότερο ευρωπαϊκό δίκτυο ε, των αρμοδίων υπηρεσιών. Αυτά λοιπόν από μένα σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Λεζερή. Ευχαριστούμε που παρουσιάσατε το έργο της Frontex. Και είναι ένα θέμα το οποίο μας μας απασχολεί ιδιαίτερα. Νομίζω ότι τώρα θα πρέπει να δώσουμε το λόγο στους συναδέλφους. Θέλω λοιπόν να συνεργαστείτε αγαπητοί συνάδελφοι όσο μπορείτε έτσι ώστε να τα πάμε καλά, γιατί έχουμε ένα τεράστιο κατάλογο, είναι τουλάχιστον 30 οι βουλευτές οι οποίοι θέλουν ε, να μιλήσουν και έχουμε λιγότερο από μία ώρα στην διάθεσή μας. Σας παρακαλήσω λοιπόν να παραμείνετε στο ένα λεπτό και επειδή ο κύριος Λεζερή μας είπε πως δεν θα είναι ε, στο γραφείο του ακόμα πολλή ώρα, θα πρότεινα στον πρώτο γύρο ερωτήσεων να θυμόμαστε πως ε, αν έχουμε κάτι να ρωτήσουμε ε, τον ε, διευθυντή της ε, Frontex, να κάνουμε την ερώτηση πρώτη. Ξέρω πως κάποιοι συντονιστές, και διορθώστε με, ο κύριος Προκατσίνη από την ECR και ο κύριος Ταρντίνο από την ID, θα ήθελα να κάνω τις ερωτήσεις του στο δεύτερο γύρο. Οπότε στον πρώτο γύρο θα τηρήσω τις ισορροπίες και θα δώσω το λόγο στους συντονιστές που το ζήτησαν. Και στο δεύτερο γύρο θα τους συμπεριλάβω και τους υπόλοιπους. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να ε, είστε όσο περισσότεροι, αλλά βοηθήστε μας με το χρόνο. Ένα λεπτό παρακαλώ. Η κυρία Ντυπού, έχετε το λόγο. Μπορώ, συγχωρέστε με. Θα ήθελα να διευκρινίσω και για μένα και για τον κύριο Προκατσίνη ότι ως εκπρόσωποι της ομάδας μας θα θέλαμε να κάνουμε ρωτή στην κυρία Ρακέτε. Αν μπορούμε να τις θέσουμε στον πρώτο γύρο, θα τις θέσουμε στον πρώτο γύρο. Ναι, φυσικά, εσείς είστε συντονιστέ των ε, πολιτικών σα ομάδων, επομένως έχετε κάθε δικαίωμα να κάνετε ό,τι ερώτηση θέλετε. Απλώς εγώ πρότεινα απλώς ότι αν υπάρχει κάτι ε, το οποίο θέλετε να απευθύνετε στο διευθυντή του Frontex, καλό να το κάνετε στον πρώτο γύρο. Ο κύριος Προκατσίνη. Ναι, πολύ καλά. Απλώς θα θέλαμε να δώσουμε τη δυνατότητα στο δεύτερο γύρο να ρωτήσουμε ε, αλλού. Ναι, φυσικά. Η κυρία Ντύπο. <clears throat> Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς ε, να ευχαριστήσω όλους τους προσκεκλημένου για τις πολύ ενδιαφέρουσε παρεμβάσει τους. Δεν ε, μπορώ να επικεντρώσω την ερώτησή μου μόνο στην Frontex. Ε, είναι βέβαια μια ερώτηση προς τον κύριο Λεζερή, αλλά και προς τους υπόλοιπου προσκεκλημένου. Ίσως ξαναπάρω το λόγο στο δεύτερο γύρο. νομίζω πως συμφωνούμε όλοι ότι η απώλεια ανθρώπινων ζωών στη Μεσόγειο πρέπει να λάβει ένα τέλος. Και αυτό νομίζω φάνηκε και από την σημερινή συζήτηση. Φάνηκε επίση και το πόσο περίπλοκο είναι το θέμα αυτό και πόσο σημαντικό και επίγον είναι να βρεθεί ένα ε, μόνιμο ε, λειτουργικό ε, βιώσιμο μηχανισμό έρευνα και διάσωση, ο οποίο θα είναι ενταγμένο στο ε, γενικότερο ευρωπαϊκό ε, σύστημα ε, ασύλου. Είναι πολύ σημαντικό για να μην χαθούν άλλε ανθρώπινε ζωέ. Αυτό όμω χρειάζεται συνεργασία με πολλούς, από πολλού φορεί, από τι χώρε προέλευση, διέλευση, από τι μη κυβερνητικέ οργανώσει, όπω ακούσαμε. Γι' αυτό λοιπόν η ερώτησή μου προ τη Frontex και προ του υπόλοιπου προσκεκλημένου είναι η εξή. Χρειαζόμαστε μεν μία μια, καταπο... μια βιώσιμη προσπάθεια καταπολέμησης της διακίνησης ανθρώπων, έτσι ώστε να μην βάζουν τη ζωή τους σε κίνδυνο διασχίζοντας τη θάλασσα, έτσι ώστε να μην εποφελούνται οι εγκληματίες. Πώς λοιπόν, μπορείτε να... Ε, πώς μπορεί, λοιπόν, προτείνετε να γίνει αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Σημειώστε παρακαλώ τις ερωτήσεις. Θα κάνουμε ένα σύντομο γύρο ερωτήσεων, σύντομο γύρο απαντήσεων και μετά θα συνεχίσουμε. Η κυρία Τσίπελ. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ συγκεκριμένη για ένα θέμα. Ε, κύριε Λεζερή, είπατε πως το καθήκον της Frontex δεν είναι μόνο ε, η διάσωση, ε, αλλά και άλλα καθήκοντα. Όταν όμως κάνετε διάσωση και είσαστε στη θάλασσα, τι κάνετε, είστε στη Μεσόγειο τη σωστή στιγμή. Γιατί όταν βλέπετε ανθρώπους να κινδυνεύουν, το εθνικό δίκαιο το διεθνέ δίκαιο ε, σα λέει πω πρέπει να του σώζετε. Είπατε όμω πω δεν μπορείτε να του προστατεύσετε αν δεν υπάρχει προηγούμενη συμφωνία για αποβίβαση. Τι σημαίνει αυτό, ότι όταν είστε στη θάλασσα και γιουσί ανθρώπους να κινδυνεύουν δεν θα τους σώσετε γιατί δεν υπάρχει προηγούμενη απόφαση για την αποβίβαση. Νομίζω ότι αυτό καταστρατηγεί το διεθνές δίκαιο. Πρέπει να τους προστατεύετε. Είτε υπάρχει προηγούμενη απόφαση αποβίβασης είτε όχι. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ιντεβέλτ. Ευχαριστώ. Πρώτα, ε, να πω στον κύριο Λεζερή πως εγώ πάντα ακούω νομικά επιχειρήματα από δικό σας, ε, τη δική πλευρά. Δεν έχουμε εντολή, δεν μπορούμε να κάνουμε το τάδε μήνυμα, δεν μπορούμε νόμιμα να κάνουμε το άλλο. Έχετε όμως διεθνεί υποχρεώσεις. Γιατί έχω αρχίσει να αποκομίζω την εντύπωση, γιατί έχουμε συζητήσει συχνά μαζί, ότι εσείς κάνετε πολιτικές επιλογές και τα κράτη-μέλη δεν αναλαμβάνουν τι ευθύνε τους. Προτιμούν να κατηγορήσουν ΜΚΟ για διάσωση στη Μεσόγειο, για παράδειγμα. Προσπαθούν να ποινικοποιήσουν τη διάσωση. Στην Ισπανία, για παράδειγμα, ακούσαμε πως εσείς ρωτάτε αυτούς που έχουν διασωθεί τι κάνουν οι ΜΚΟ, γιατί, γιατί είχε το σκοπό να ποινικοποιήσετε τη δράση τους. Μου δώσετε δύο μου εξηγήσει για τα θέματα αυτά επίσης, για τα όσα συζητήσαμε την περασμένη φορά, για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η κατανομή ε, και, και το πώς μοιράζεται τις πληροφορίες. Δηλαδή κινδυνεύει κάθε σκάφος. Την περασμένη φορά μας είπατε ότι γίνεται μέσω του κέντρου ε, διάσωσης που στέλνει τις πληροφορίες και εμείς μετά ε, μοιράζουμε τις πληροφορίες σε άλλους. Εγώ νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνεται άμεσα. Ε, δηλαδή αν υπάρχουν μη, σκάφη μήκη όπου στην περιοχή πρέπει αμέσως να ενημερώνονται. Και ποια είναι η διαδικασία ε, εντολής ε, το σκάφος που διασώζει δεν θα πρέπει να ακολουθεί ε, τις επιθυμίες του κράτους, του κράτους μέλους. Εσείς εκπροσωπείτε την Ευρωπαϊκή Ένωση και το κατά πόσο θα ποινικοποιηθεί η δράση κάποιων ΜΚΟ είναι εθνικό θέμα και όχι δική σας απόφαση. Σας παρακαλώ πολύ ένα λεπτό. Ένα λεπτό γιατί ο κατάλογος είναι όλο και πιο γεμάτος. Για τους πράσινους ο κύριος Μάρκαρτ είναι ο πρώτος ομιλητής. Κυρία Τρίκ, κυρία Στρίκ παρακαλώ. Πριν από 7 χρόνια παρουσίασα εδώ στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ την έκθεσή μου για τις ζωές που χάνονται στη Μεσόγειο εκ μέρους του Συμβουλίου της Ευρώπης. Και τότε είχαμε πει πως 70 άτομα αφέθηκαν στην τύχη τους στη Μεσόγειο και περισσότεροι ε, έχασαν τη ζωή τους και ζήτησαν να υπάρξει ένα σύμφωνο για τη Μεσόγειο για να μην υπάρχει κανένα κενό υπευθυνότητα. Και έκτοτε Εχάθηκαν πάρα πολλές ζωές και θα ήθελα να ευχαριστήσω τις οργανώσεις και τα κράτη-μέλη που έχουν σώσει ανθρώπους και πιο συγκεκριμένα την Sea-Watch και την κυρία Ρακέτε. Τώρα έχουμε και κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις. το τόπος ασφαλής, τι σημαίνει αυτό, γίνεται αποβίβαση στη Λιβύ. Είναι ασφαλή η Λιβύη. Νομίζω το ξέρουμε όλοι ότι είναι ασφαλή. Δεν μπορούμε να το συμπεριλάβουμε, αλλά θέλω αυτό να μου το επιβεβαιώσετε. Επίση, η ύπατη αρμοστία ήδη είπε πως πριν από δύο μήνες δεν μπορούμε να θεωρούμε πως η Λιβική ακτοφυλακή μπορεί να διαχειριστεί όλες τις επιχειρήσεις διάσωσης. Γιατί η απόκρισή τους είναι ε, στο επίπεδο διάσωσης και έρευνας εξαιρετικά απρόβλεπτη. Μήπως μπορείτε να το σχολιάσετε αυτό, κύριε Τασάρα. Και επίσης η MRCC ε, Ρώμης συντονίζει το κομμάτι που είναι στην Τρίπολη της Λιβύης. Τι σημαίνει αυτό και τι γίνεται με τις ε, παραβιάσεις ε, που κάνει η Λιβική Ακτοφυλακή. Ποιος είναι υπεύθυνο, η MSSR Ρώμης. Τι μπορείτε να πείτε εσείς και συγκεκριμένα στη Frontex δεν έχετε σκάφη, έχετε μόνο αεροπορική ε, παρακολούθηση. Ε, το άρθρο ο, αυτό της Άγκλος δεν σημαίνει ότι καλύπτονται και τα αεροπορικά μέσα και θα πρέπει και αυτά αμέσως να παρέχουν ε, διάσωση. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, βοηθήστε με, είμαστε πάρα πολύ. Μην μιλάτε πάνω από ένα λεπτό. Και αν περάσουμε το χρόνο μας, δεν θα έχουμε διερμηνία. Βοηθήστε με να σας βοηθήσω. Θέλετε το χρόνο σας, ε, κυρία Ταρντίνο, εκ μέρους του ID. Κύριε Πρόεδρε, εγώ φοβάμαι ότι μετά δεν θα υπάρχει χρόνος, επομένως θα θέσω τώρα την ερώτησή μου στην κυρία Ρακέτε. Από ό,τι φαίνεται, χάρη σε εσά έφτασαν στην ε, Ιταλία τρει βασανιστέ και βιαστέ από τη Συρία, που φαίνεται ότι έχουν διαπράξει πονίδα στα εγκλήματα στο σκάφο που χρησιμοποιήσετε εσεί για να κάνετε μια πολιτική μάχη κατά του Ματέο Σαμβίλη και τη Ιταλία και όχι μια ανθρωπιστική αποστολή. Αυτό είναι το ίδιο το οποίο επέτρεψε να μαζέψετε και στα μέσα μαζική δικτύωση πάνω από 300.000 ευρώ. Το γνωρίζετε ότι μεταφέρετε αυτού του ανθρώπου, γιατί αυτό θα ήταν όντω στρέβον παράγοντο η δικαιοσύνη στην οποία αναφερθήκατε προηγουμένω. Έχετε συνειδητά παραβιάσει την Ιταλική νομοθεσία, θέσατε σε κίνδυνο τη ζωή ανθρώπων εν στολών, καθώ επίση και των ανθρώπων επί του σκάφου, που κανένα από αυτού δεν είχε ενδείξει βασανισμών ή κάποιων σοβαρών ασθενειών. Στην πραγματικότητα, εμεί είμαστε αυτοί που είμαστε απαγορετευμένοι από αυτή την Ευρώπη που υποδέχεται στην, ε, στο σπίτι των τίμιων Ευρωπαίων ανθρώπων εσά σαν να είστε ηρωίδε. Εσεί που θα έπρεπε να ε, διδάξετε υποτίθεται σε ένα καθολικό και φιλόξενο λαό όπως η Ιταλία πώς θα έπρεπε να υποδέχεται ανθρώπους. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Προκατσίνη, ένα λεπτό παρακαλώ. Ναι, πολύ σύντομα. Προφανέ κανένα δεν θέλει να ποινικοποιήσει τι δραστηριότητε διάσωση στη θάλασσα. Ε, την οποία άλλωστε κάνει με ιδιαίτερο ε, ε, ικανό τρόπο η Ιταλική Ακτοφυλακή, την οποία ευχαριστώ γιατί το κάνει και μακριά από τις τηλεοπτικές ε, κάμερες. Το πρόβλημα είναι η συνεργασία με τους διακινητές, με την παράνομη μετανάστευση και με την διακίνηση ανθρώπων. Και η ερώτησή μου, την οποία θα ήθελα να απευθύνω στο διευθυντή του Frontex, είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Αν δούμε τα στατιστικά στοιχεία, εμείς γνωρίζουμε ότι φέτος το 2019 σε σχέση με το 2019 οι νεκροί στη θάλασσα μειώθηκαν από 2.818 στους 929, δηλαδή πάνω από τους μισούς. Ε, παρά το γεγονός βέβαια ότι μια ζωή στη θάλασσα είναι τραγωδία ούτως ή άλλως, ε, πώς ε, εξηγείται το γεγονός ότι το τελευταίο έτος ε, μειώθηκαν στο ίμιση οι θάνατοι στη θάλασσα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Από ό,τι κατάλαβα από την ΚΟΕ θα μιλήσει η κυρία Μπιόρκα. Α, η κυρία Έρνστ. Ε, ε, Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα λοιπόν να πάρω μια απόσταση από τους δύο προλαλήσαντες, να το πούμε αυτό. Κυρία Ρακέτα, έχω μια ερώτηση για εσάς. Σε αυτές τις μέρες που μείνατε στη θάλασσα, τι έγινε. Προσπαθήσατε να έρθετε σε επαφή με την Ιταλική ακτοφυλακή έτσι ώστε να σας βοηθήσουν το συντομότερο. Ε, ποιες ήταν οι ενέργειες που κάνατε και τι διαδραματίστηκε, πώς εκτελήθηκαν τα γεγονότα. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ήθελα να μου πείτε ποιες ενέργειες έχετε κάνει στο πλαίσιο των συνομιλιών σας με τα κράτη-μέλη έτσι ώστε ε, να σταματήσει η ποινικοποίηση των μη κυβερνητικών οργανώσεων που αναλαμβάνουν τέτοιες επιχειρήσεις. Έχετε διοργανώσει κάποιο συνέδριο. Τι κάνετε για αυτό το πράγμα ή τι έχετε ήδη κάνει. Και ε, άλλη μια ερώτηση για όλους. Η Λιβύη ε, χαρακτηρίζεται ως ασφαλή, σε τρίτη ε, χώρα. Εγώ θα ήθελα να μου πείτε εάν έστω και ένας από εσά θεωρεί τη Λιβύη ασφαλή χώρα. Μα έχετε πει πως θα μας δοθούν επιπλέον 15 λεπτά διερμηνίας. Αλλά μετά θα φύγουν οι διερμηνείς και θα πρέπει να μιλάμε αγγλικά. Προτείνω λοιπόν πρώτα να απαντήσει ο κύριος Λεζερή για τρία λεπτά και μετά το υπόλοιπο πάνελ. Και μετά δεύτερος γύρος ερωτήσεων. Κύριε Λεζερή, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ ε, και όλους όσους υποβάλατε ερωτήσεις. Επιβεβαιώνω Είμαστε παρόντες στην Κεντρική Μεσόγειο με σκάφη στα πλαίσια της επιχείρησης Θέμης στην επιχειρησιακή περιοχή που επιβλέπει. Και επίσης έχουμε και αεροσκάφη τα οποία κάνουν περιπολίες στην Κεντρική Μεσόγειο. Όχι ως τμήμα της επιχειρήσεως Θέμης, Άρα στα πλαίσια της Eurostore, το οποίο σημαίνει ότι περιπολούμε με τα δικά μας σκάφη, αεροσκάφη και μόλις βρούμε περιστατικό ή κατάσταση ενδεχόμενης ή πραγματικής διάσωσης και έρευνας, μοιραζόμαστε τις ε, πληροφορίες με τα Εθνικά Θαλάσσια Κέντρα Συντονισμού. Άλλες φορές βλέπουμε και άλλα περιστατικά που δεν έχουν να κάνουν με έρευνα και διάσωση, αλλά περισσότερο με ε, έργο διοκτικών αρχών Πάντω εμεί, σε πραγματικό χρόνο στέλνουμε τι πληροφορίε. Για την έρευνα και διάσωση, να σα πω το εξή, πω σε αυτές τι περιπτώσει μοιραζόμαστε με όλα τα κέντρα συντονισμού, θαλάσσιου συντονισμού τη περιοχή, μοιραζόμαστε τι πληροφορίε σύμφωνα με το θαλάσσιο δίκαιο και δεν είμαστε υποκείμενοι σε οποιαδήποτε πολιτική επιρροή όταν υπάρχει περίπτωση έρευνα και διάσωση επιτακτική ανάγκη. Γιατί αυτό τότε πρέπει να συμβεί και η επιχειρησιακή απόκριση δίδεται. Δεν μπορούμε όμως να είμαστε εμείς ο συντονιστής σε αυτές τις δράσεις. Γιατί δεν έχουμε τέτοια εντολή. Και όταν εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση Όταν λοιπόν είμαστε δραστήριοι σε περιοχές ε, που είναι ε, εθνικής κυριαρχίας, και επειδή οι εθνικοί νομοθέτε δεν έχουν δώσει υπερεθνικές αρμοδιότητε σε ευρωπαϊκέ υπηρεσίες, δεν είμαστε σε θέση να αναλάβουμε δραστηριότητα, πρωτοβουλία και να δράσουμε ανεξάρτητα, αλλά πρέπει να ακολουθήσουμε τι οδηγίε, οι οποίε μα δίδονται στα πλαίσια του ε, τακτικού ε, επιχειρησιακού σχεδιασμού. Και αυτό για να ε, απαντήσω στις ερωτήσει των ε, ευρωβουλευτών. Έχουμε επιχειρησιακό σχέδιο και είναι δικό μα καθήκον να εξασφαλίσουμε πω το επιχειρησιακό σχέδιο δεν ευθυγραμμίζεται μόνο με την εντολή μας, αλλά παράλληλα και με τις βέλτιστες πρακτικές, οι οποίες σχετίζονται όχι μόνο με την επιτήρηση των συνόρων, αλλά και με το έργο των διοκτικών αρχών και παράλληλα είναι σε θέση να θέσουν σε εφαρμογή τις βέλτιστες πρακτικές για τις δράσει έρευνα και διάσωση. Για το πώ μπορώ να εξηγήσω τον αριθμό των ε, θυμάτων και το γιατί μειώθηκε αυτός το βλέπω σε συνδυασμό με, το, με τη μείωση των ανθρώπων οι οποίοι προσπαθούν να περάσουν αυτή τη θάλασσα, μείον 80% πέρσι, Μείωνο 80% στην κεντρική Μεσόγειο. Uh, of of, uh, of... Και αυτό σίγουρα εξηγεί γιατί μειώθηκαν και τα θανατηφόρα περιστακτικά. Σημαντικό επίσης είναι να μπορούμε να πατάξουμε τα εγκληματικά δίκτυα, γιατί και αυτά είναι παρόντα σε τρίτες χώρες, δεν είναι όλα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να ε, συνεργαστούμε μαζί τους μπορούμε εμείς να συλλέξουμε και να διεκπαιρεώσουμε ε, στοιχεία που θα τροφοδοτήσουν τις έρευνες της Europol ή των Εθνικών Διοκτικών Αρχών. Αυτό είναι καθήκον μας γιατί είμαστε και εμείς διοκτικό όργανο και με τον τρόπο αυτό μπορούμε να πατάξουμε το διασυνοριακό έγκλημα, το τράφικινγκ και αυτό είναι καθήκον καθημερινού για οποιαδήποτε προσπάθεια έρευνας και διάσωσης την οποία συντονίζουμε είτε ε, με τους θαλάσσιους πόρους που έχουμε είτε μέσω των ε, ε, είτε μέσω των αεροπλάνων μας, τα οποία μπορούν να είναι αεροσκάφη ή drones. Ε, ευχαριστώ πολύ. Είναι δύσκολο το καθήκον μου και ήταν και καλή προσπάθεια Μα δεν απάντησε. Δεν απάντησε την ερώτηση που έκανα. Η Λίβη είναι ασφαλής τόπος, είναι ασφαλής χώρα, πείτε μου. Ναι. Θέλετε, θέλετε να το απαντήσετε αυτό. Ευχαριστώ. Υποθέτω όπως ως εκτελεστικός διευθυντής υπηρεσίας δεν μπορώ να αποφανθώ εγώ αν κάποια χώρα είναι ασφαλής ή όχι. Εγώ ποτέ δεν είπα πως η Λιβύη είναι ασφαλής χώρα πάντως. Αυτή είναι η κανόνα του παιχνιδιού. Έχουμε βίντεο link, ο χρόνος είναι περιορισμένος. Ας ακούσουμε και τους υπόλοιπους στο πάνελ. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για όλες προσπάθειες που έχετε κάνει και θα κάνετε, παρακαλώ πολύ, εσείς πρώτος και μετά οι υπόλοιποι. Έτσι ώστε οι ευρωβουλευτές να κάνουν και άλλες ερωτήσεις μετά. Well, Σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχά, νομίζω πω πρέπει όλοι να αναγνωρίσουμε το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Frontex στη διάσωση ανθρώπινων ζωών μέσω των επιχειρήσεών τη. Πράγματι έχετε σώσει πολλές ζωές. Όμως, ε, σχετικά με το αν η Λιβύη μπορεί να θεωρηθεί ασφαλής ε, τόπος, νομίζω πως ε, όχι, δεν μπορεί να θεωρηθεί ασφαλής χώρα. Γι' αυτό λοιπόν και η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιεί σκάφη για να διεξαγεί αυτές τις επιχειρήσεις αποβίβασης. Επίσης πρέπει να τονίσω ότι η απάντηση για αυτό που συμβαίνει στη Μεσόγειο αυτή τη στιγμή δεν είναι τόσο εύκολη. Είναι, πρέπει να είναι κομμάτι μιας ευρύτερη στρατηγικής, μιας ε, πιο συνολικής ολιστικής προσέγγισης. Και χρειάζεται να βρεθούν απαντήσεις και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και από τα κράτη-μέλη, έτσι ώστε να βρούμε μια σταθερή λύση. Σταθερή, αλλά όχι μόνο ε, για τις επιχείρησεις αλλά και για τη συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Χρειάζεται λοιπόν ε, να δούμε τι γίνεται εκεί αλλά και να αναγνωρίσουμε ότι έχουν γίνει πολύ θετικές ενέργειες ε, τώρα πρόσφατα στη Μάλτα. Χρειάζονται όμως πολλά περισσότερα έτσι ώστε να βρούμε λύση για το ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου και για διάφορα οριζόντια θέματα, μεταξύ άλλων και την καταπολέμηση ε, της διακίνησης ανθρώπων και του λαθρεμπορίου. Δεν πρέπει να εθελοτυφλούμε μπροστά σε αυτά που πηγαίνουν. Αυτό, είναι, αυτό που γίνεται με την διακίνηση ανθρώπων είναι επιχειρήσει ε, κανονικότατες, επιχειρηματικό μοντέλο αυτών των εγκληματικών οργανώσεων. Μπορούμε να διοργανώσουμε διάφορες ημερίδες ε, για την ανθρωπιστική βοήθεια και για τη θέση της ε, μας. Ποια είναι η θέση μας τώρα. Εμείς ε, κάναμε μία αξιολόγηση το 2017 όπου υπήρξαν αρκετά ευρήματα και αποδεχόμαστε ότι δεν υπάρχει αρκετή σαφήνεια. Ε, εκφράσαμε τις ε, μεγάλες μας ανησυχίες και την ανάγκη που υπάρχει για έλεγχο και παρακολούθηση. Ζητήσαμε λοιπόν τη συνδρομή όλων των ενδιαφερόμενων φορέων και να είστε σίγουροι πως έχουμε ανοιχτό μυαλό σε ό,τι αφορά τα θέματα αυτά. Ελπίζω το νέο Σώμα των Επιτρόπων να ασχοληθεί με το θέμα αυτό και να εξετάσει τις ε, δυνατότητες που έχουμε αντιμετώπισης του προβλήματος. Αυτά από την δική δική μου μεριά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος στον κύριο Μόλναρ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για το λόγο. Καταρχάς θα ήθελα να απαντήσω στην ερώτηση της κυρία Στρίκ. Δεδομένου ότι η Λιβύη δεν ανταποκρίνεται στις ε, εκκλήσεις για βοήθεια. Νομίζω ότι η Επιτροπή για την ε, Ασφάλεια στη Θάλασσα μπορεί να δώσει ορισμένες ε, κατευθυντήριες γραμμές και ορισμένες οδηγίες για το πώς μπορεί να διεξαχθεί μια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Όταν κάποιο κράτος δεν μπορεί ή δεν θέλει να αναλάβει τις ευθύνες του. Θα πρέπει λοιπόν οι ευθύνες να μεταβούν στον επόμενο, στην αλυσίδα. Έτσι ερμηνεύουμε εμείς ε, το νόμο. Το άρθρο 98 της ε, UNCLOS σχετικά με, τα, ε, με τη διάσωση με αεροσκάφος τεχνικά δεν είναι δυνατόν λόγω του δικαίου της θάλασσας, λόγω των ορισμών ενός σκάφους Υπάρχει όμως ένα εγχειρίδιο για την έρευνα και διάσωση στη θάλασσα, το οποίο καλύπτει και περιπτώσεις αεροσκαφών τα οποία διεξάγουν πτήσεις ε, παρακολούθησης. Αυτό τώρα, εάν θα μπορέσει να εφαρμοστεί και στις ε, περιπτώσεις ε, ανάπτυξης αεροπορικών δυνάμεων, θα το δούμε. Θα ακολουθήσει μία εκτίμηση αντικτύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όμως ε, αυτό δεν ε, είμαστε ε, αρμόδιοι να το αποφασίσουμε μόνοι μας. Κύρια Ρακέτε, έχετε το λόγο να απαντήσετε στις ερωτήσεις από την καρδιά σας. Σας παρακαλώ να είστε σύντομοι για να ακολουθήσει και η επόμενη συζήτηση. Νομίζω ότι έγινε σαφές εδώ από πολλούς στο πάνελ μέχρι τώρα πως η διάσωση ανθρώπων στη θάλασσα είναι διεθνής υποχρέωση. Εγώ προσωπικά δεν αντιλαμβάνομαι πώς μπορεί η Ιταλική χώρα να περνά εθνικό νόμο ο οποίος δεν είναι σύμμορφος με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Και είδαμε ότι μετά από τη σύλληψή μου ο δικαστή στην Ιταλία, στο Αγκριτζέντο, σαφέστατα αποφάνθηκε ότι είχα ακολουθήσει την υποχρέωση να διασώσω και οτιδήποτε συνέβη συμμορφούταν πλήρως προς το δίκαιο της θάλασσας. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη που ε, ανησυχείτε για τους βασανισμούς στη Λιβύη, γιατί εγώ προσωπικά ανησυχώ πάρα πολύ Πρέ... Συναντούμε ανθρώπους ε, οι οποίοι βασανίζονταν σε καθημερινή βάση στα σκάφη ε, στη θάλασσα. Και φυσικά ε, όταν προσπαθούμε να διασώσουμε κάποιον, δεν γνωρίζουμε και την ιστορία του. Αν σας ανησυχούν όμως οι βασανισμοί στη Λιβύη πραγματικά, τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να σταματήσει κάθε συνεργασία με τη Λιβυκή Ακτοφυλακή, η οποία συνεχώς παίρνει ανθρώπους από τα διεθνή ύδατα και τα ξαναπηγαίνει σε αυτά τα κέντρα κράτησης, ε, σε αυτούς τους ανθρώπους που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτοί είναι γνωστοί και αυτούς προσπαθούν, από αυτούς προσπαθούν να ξεφύγουν αυτοί οι άνθρωποι. Και κάτι ακόμα το οποίο θα ήθελα να προσθέσω, πολύ σύντομα. Ισχύει επίσης ότι τα διάφορα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποστηρίζουν διαφορετικές ομάδες στον εμφύλιο πόλεμο στη Λιβύη και παρατείνεται έτσι αυτός ο πόλεμος και δημιουργεί μια κατάσταση στην οποία μπορούν να υπάρχουν τέτοιες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Πλήρχε Σάρα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να απαντήσω στην κυρία Στρίκ. Η Ιταλική εκτοφυλακή, καταρχάς, εδώ και χρόνια τηρεί όλη τη διεθνή νομοθεσία η οποία κυρώθηκε με νόμο του Ιταλικού κράτους. Ε, αυτό λοιπόν ε, μας οδήγησε στη διάσωση ε, χιλιάδων μεταναστών στη διάρκεια των ετών, αλλά ε, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η ίδια νομοθεσία, η οποία επαναλαμβάνω κυρώθηκε μέσω νόμου, προβλέπει ότι όταν υπάρχει ένα κέντρο διάσωσης ε, το οποίο είναι υπεύθυνο για κάποια περιοχή, το πρώτο κέντρο διάσωσης που λαμβάνει ε, την ε, SOS ε, πρέπει να κάνει τις πρώτες δραστηριότητες αλλά πρέπει να ενημερώσει και το κέντρο το οποίο είναι υπεύθυνο αναπεριοχή γιατί από εκεί και πέρα αφού γίνουν οι πρώτες ενέργειες είναι υπεύθυνο αυτό το κέντρο. Στο παρελθόν δεν είχαμε συνομιλητές αλλά εξ όσων αφορά αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία αναγνωρίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη. Υπάρχει ένα κέντρο διάσωση στη Λιβύη. Η Λιβική ακτοφυλακή έχει επιχειρησιακέ δυνατότητε οι οποίε αυξήθηκαν. Επομένω, εμεί, επειδή πάντα τηρούμε την νομοθεσία, διεθνή νομοθεσία και εθνική νομοθεσία, επαναλαμβάνω, πρέπει απόλυτα να ενημερώσουμε το κέντρο το οποίο είναι αρμόδιο για την περιοχή. Αλλιώ ε, παρανομούμε εμεί. Εμείς λοιπόν ερχόμαστε σε επαφή μαζί του. το κέντρο της Λιβύη αναλαμβάνει τον συντονισμό και γίνεται υπεύθυνο για την ε, δράση διάσωση στη θάλασσα. Κατά τα άλλα η Ιταλία ποτέ δεν έχει αποχωρήσει από οποιαδήποτε επιχείρηση διάσωσης σε οποιαδήποτε περιοχή εκτός από τα ε, ύδατα της δική της ευθύνη στη Μεσόγειο. Έχουμε συντονίσει ακόμα και επιχειρήσεις διάσωσης στον Ειρηνικό ωκεανό και στον Ατλαντικό ωκεανό ως ε, πρώτο κέντρο διάσωσης που λαμβάνει το σήμα εκτάκτου ανάγκης. Ε, μετά, εάν δεν γίνει μεταβίβαση στο αρμόδιο ε, κέντρο διάσωσης, προβλέπεται ότι η ευθύνη παραμένει του πρώτου κέντρου. Αυτό και βάσει τη σύμβαση ΣΑΡ και βάσει τη σύμβαση του Αμβούργου κλπ. Εμεί δεν έχουμε επαναχωρήσει ποτέ, αλλά πρέπει να τηρούμε τη διεθνή και εθνική νομοθεσία, επαναλαμβάνω. Εμεί ευχαριστούμε, τα Σάρα. Τώρα, είναι 11 παρατέταρτο. Προβλεπόταν η συνεδρίασή μα μέχρι τι 11. Θα μείνουμε μέχρι τι 11 και 4 και θα υπάρξει χρόνος για όλα τα, κράτη μέλη, για όλα τα μέλη συγγνώμη, να μιλήσουν μέχρι 30 άτομα, αλλά από τις 11 και 4 και μετά πρέπει να μιλάμε όλοι στα αγγλικά. Αυτό είναι ο κανόνα, γιατί θα σταματήσει η διερμηνία. Ακόμα και τα μέλη του πάνελ θα πρέπει να απαντήσουν στα αγγλικά, γιατί η διερμηνία θα αποχωρήσει. Ένα λεπτό παρακαλώ, ώστε να μπορέσετε όλοι να πάρετε το λόγο. Ξεκινάμε με την κυρία Στάτλερ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω το εξή, πως είναι μια ανθρώπινη καταστροφή, είναι ανθρώπινες τύχες και γι' αυτό το σύστημα που θα επιλέξουμε θα πρέπει να λειτουργεί και δεν θα πρέπει να αφήνονται στην τύχη τους και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε πως η λειτουργία θα είναι η απαραίτητη. Δεν θα χωριστούμε σε καλούς και κακούς, καλά κράτη και κακά κράτη. Είναι ένα ανθρώπινο, ευρωπαϊκό, διεθνέ, καθήκον και έχει να κάνει με το να σώσουμε ζωέ και δεν θα πρέπει να επιτρέπουμε το τράφικινγκ, θα πρέπει με έναν τρόπο να το ε, πατάξουμε και σε μια ιστορική στιγμή η καινούργια πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε στη μεταναστευτική πολιτική θα ξεκινήσουμε από μηδενική βάση και θα λάβουμε υπόψη όλε τι διαστάσει τι οποίε ε, ανέφεραν εδώ οι διάφοροι ε, ομιλητές. Έχουμε τη Frontex, έχουμε τη συνεργασία, αλλά χρειάζεται και ένταξη των ανθρώπων αυτών. Ένταξη όσων μένουν στις χώρες μας. Και γι' αυτό σας ρωτώ, Πώς πρόκειται να γίνει αυτή η αλλαγή. Δεν βλέπετε να υπάρχει πρόβλημα το ότι είμαστε ελκυστικοί. Ο κύριος Μωράης. Όταν θέλουμε λοιπόν να σταματήσουμε την ποινικοποίηση της δράσης ανατόμων και ΜΚΟ, αυτό το οποίο έχουμε κάνει είναι ε, με ποιο τρόπο. Κύριε Σάτερ, πείτε μας πώς μπορούν να σας βοηθήσει η καινούργια Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είπαμε νομική υποχρέωση, αλλά οκτώ κράτη-μέλη μόνο έχουν αποποινικοποιήσει το θέμα της αλληλεγγύης. Άρα λοιπόν η νέη Επιτροπή, και το είπαμε και με την νέα αρμόδια Επίτροπο, πώς θα αντιμετωπίσει το θέμα της δίωξης όσων κάνουν διάσωση ε, και τι γίνεται με την ρήτρα εξαίρεσης ε, και απαλλαγή ευθύνη στη συγκεκριμένη περίπτωση. Γιατί τα όσα είδαμε πέρσι μας υπέδειξαν πως η Λιβύη δεν είναι ασφαλής χώρας και θα ήθελα κι εγώ ε, να, να ξεχωρίσω τη θέση μου από σχόλια προηγουμένων συναδέλφων. Ε, κυρία Κλέρ, έχω την εξή ερώτηση. Λέει η κυρία Κέλλερ, Όπω και ο κύριος Μοράλε Μωράης, θέλω να ρωτήσω το εξή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναθεωρήσει την, διαδικασία, την ε, οδηγία διευκόλυνσης, θα δώσει κατευθυντήριες γραμμές, θα βάλει στόχους, έτσι ώστε να μην ποινικοποιούμε πλέον άτομα ή οργανώσεις οι οποίες βοηθάνε βοηθάνε, προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια και διευκολύνουν την πρόσβαση. Και θα ήθελα να εκφράσω ε, και τον θαυμασμό μου προς την κυρία Ρακέτη. Ε, Κυρία Ρακέτε, ήθελα να πω το εξής. Εσείς φέρατε ένα σκάφος ολόκληρο παράνομων μεταναστών σε Ιταλικό λιμάνι. Τρεις εγκληματίες οι οποίοι ε, ηγούν των ε, εγκληματικού στρατοπέδου στη Λιβύη που είχαν κατηγορηθεί για βιασμούς, για δολοφονίες, για βασανιστήρια. Αυτούς φέρατε. Μπορείτε να είστε υπέρ της μετανάστευσης, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει σε ένα νόμιμο πλαίσιο, σύμφωνα με το κοινοβουλευτικό ε, δίκαιο. Εσείς επιλέξατε το νόμο της βίας και δεν σέβεστε το γεγονός ε, πως αυτό σας έχει καταστήσει τμήμα ενός εγκληματικού δικαίου ε, που ασχολείται με το ανθρώπινο τράφικινγκ. Δεν θα έπρεπε να σας εδώ σε κελί θα έπρεπε να σας έχουν κλείσει. Ρωτώ το εξή. Πιστεύετε εσείς πως χωρίς κλειστά σύνορα ε, θα συνεχίσει ο κόσμος να έρχεται. Uh, uh, Μία ερώτηση για την κυρία Ρακέτ. Κυρία Ρακέτ, εσείς είστε εκεί στη Μεσόγειο και σώζετε ζωής και τους βοηθάτε ε, τους ανθρώπους αυτούς να περάσουν ε, στην ε, γη της επαγγελίας. Και κερδίζουν χρήματα από αυτά όσοι ε, κάνουν ε, τράφικινγκ παιδιών. Χάθηκαν ζωές ε, λόγω αυτής της προσπάθειας. Αυτό έχει συνέπειες. Συνέπειες τεράστιες. Και συμβαίνει να έρχονται άνθρωποι στη χώρα μας χωρίς καμία στρατηγική να αντιμετωπιστούν με κανένα κέρδος παρά μόνο για τους ε, διακινητές. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο για να αντιμετωπίσουμε την έκρηξη ε, στις γεννήσεις της χώρες αυτές. Αυτό θα πρέπει να είναι το μέλημά μας, όχι κάτι διαφορετικό. Thank you. I must say that I'm a little bit shocked. Με σοκάρει ο απερίφραστος ρατσισμός που εκφράστηκε εδώ σήμερα και ίσως θα πρέπει να αναλάβουμε δράση, κύριε Πρόεδρε. Να πω μόνο πως δεν μπορούμε να έχουμε μια ε, κατάσταση με αυτήν την οποία περιέγραψε η κυρία Ρακέτε, όπου αυτοί οι οποίοι σώζουν ζωέ ποινικοποιούνται και διώκονται. Θα έπρεπε να ποινικοποιούμε ε, την ε, δίωξη και την παρενόχληση αυτών. Λοιπόν, οι απαντήσει σας δεν είναι αρκετέ. Ε, ε, πώς μπορεί να βελτιωθούν τα πράγματα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. πώ θα διώξουμε και θα ποινικοποιήσουμε αυτού οι οποίοι διώκουν όσου σώζουν ζωέ. Και επίση, Frontex. Αλλά μπορεί να απαντήσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Λιβύη δεν είναι ασφαλές καταφύγιο. Γιατί λοιπόν, σύμφωνα με την επιστολή του Μαρτίου, η Frontex να δίδει πληροφορίες στην, ε, στο κέντρο διάσωσης ε, ε, της Λιβύης, το οποίο ουσιαστικά είναι pushback μέσω αντιπροσώπου. Κύριε Ούλρικ. Mr. Ulrich, please. One minute. Για ένα λεπτό. Αγαπητέ, αγαπητοί συνάδελφοι, σας άκουσα σας άκουσα για του λαθρομετανάστες που έρχονται στην Ευρώπη. Νομίζω ότι εσεί και οι διακινητές δεν διαφέρετε, γιατί ουσιαστικά εισάγετε λαθρεία ανθρώπου στην Ευρώπη. Εγκληματίες, δολοφόνους και αυτό αντίθετα με τη βούληση των κρατών μελών. Ποια είναι η διαφορά σας με τους διακίνητέ. ότι εσά σα πληρώνουν ΜΚΟ. Κυρία Ρακέτε, δεν θα μας διδάξετε εσείς ε, ποιο είναι το ιστορικό και ο καθήκον μας προς την Αφρική. Εμείς στη Σλοβακία δεν φταίμε. Θέλετε να βοηθήσετε την Αφρική, πηγαίνετε εσείς στην Αφρική. Αφήστε την Ευρώπη ήσυχη και ελεύθερη από τη δική σας παράνομη ε, οργάνωση ε, και λαθροδραστηριότητα. Θέλουμε κράτος δικαίου. Και εγώ συμφωνώ με τον κύριο Σαλβίνη. Έπρεπε να έχετε φυλακιστεί. Είστε εγκληματίας. Δεν θα έπρεπε να κάθεστε εδώ στο κοινοβούλιο.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 κύριο ε, Μόλναρ είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με όλου του ε, οργανισμού ε, δεσμεύονται από το άρθρο 98, όμω οι επιπτώσει στην πράξη δεν είναι και τόσο σαφείς. Αν η Frontex έχει πληροφορία ότι υπάρχουν άνθρωποι που κινδυνεύουν στη θάλασσα, δεν καθιστά αυτό υποχρέωση να ενημερώσουν τα σκάφη που βρίσκονται κοντά ότι υπάρχουν άνθρωποι που κινδυνεύουν. Δεν είναι υποχρέωση της Frontex, ναι ή όχι. κύριος Μπαρτόλο. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, το ήξερα. Εγώ είχα ετοιμάσει μια παρέμβαση, αλλά είμαι υποχρεωμένος να αποστασιοποιηθώ πλήρως από αυτό που είπαν οι Ιταλοί συνάδελφοι, οι οποίοι ανήκουν στη Λέγκα και επέτρεψαν να περάσουν κάποια ε, διατάγματα νόμου τα οποία ε, έκαναν παράνομη τη διάσωση ανθρώπων. Και πραγματικά ντράπηκα. Ντράπηκα. Ε, Αντιθέτω, είμαι ιδιαίτερα περήφανο για την ακτοφυλακή, που εδώ και 30 χρόνια συνεργαστήκαμε και διέσωσαν χιλιάδε ανθρώπου. Αυτή είναι η Ιταλία. Δεν είναι αυτή του Σαλβίνη. Και να πω σήμερα, που είναι η μέρα μνήμη, είναι 3 Οκτωβρίου, είναι ημέρα στην οποία εγώ στις 3 Οκτωβρίου του 2013 ήμουνα στην Λαμπεντούζα. 30 χρόνια ήμουν γιατρός στη Λαμπεντούζα και έσωζα αυτούς του ανθρώπους. 360 άνθρωποι πέθαναν λίγα ε, χιλιόμετρα από την ακτή και πραγματικά εκείνη την ημέρα δεν ήξερα τι να πω και είναι συμβολικό να βρισκόμαστε εδώ και να μιλάμε για έρευνα και διάσωση αυτή την ημέρα. Η τραγωδία αυτή είναι ένα από του λόγου για του οποίου βρίσκομαι εδώ σήμερα. Άφησα τη δουλειά μου που την αγαπώ πάρα πολύ και η απάντησή μου ή μάλλον η ερώτησή μου την έθεσε ο Κλοντ Μωρά. Αλλά πραγματικά ένιωσα την υποχρέωση να αποστασιοποιηθώ πλήρως από αυτά τα οποία ακούστηκαν ε, για την κυρία Ρακέτα, που είναι η πραγματική πλήρχος. Αυτή είναι η πραγματική πλήρχο. Ευχαριστώ πολύ. Regarding this point... Σε ό,τι αφορά αυτό που μόλις είπατε, κύριε Μπαρτόλο, πρέπει να πω ότι έχετε κάνει μια πολιτική δήλωση. Έχετε εκθέσει τις απόψεις σας για αυτό το ζήτημα, όμως νομικά πρέπει να προσθέσω και κάτι άλλο. Στο πλαίσιο της ελευθερίας ε, της έκφρασης των ε, εκλεγμένων αντιπροσώπων λοιπόν εδώ που έχουν εκλεγεί δημοκρατικά. Δεν υπάρχει κανένα νόμο δικαίωμα δυσφήμισης. Οι προσκεκλημένοι που βρίσκονται στο πάνελ, σε αυτήν την ακρόαση, ε, είναι άνθρωποι ε, τους οποίους δεν έχετε κανένα δικαίωμα να δυσφημείτε και να προσβάλλετε σε αυτήν εδώ την Επιτροπή. Έχετε λοιπόν απόλυτο δίκιο, κύριε Μπαρτόλο. move... Περνάμε τώρα στον κύριο Μάρκαντ από τους Πράσινους. Νομίζω πως ε, δεν έχει μείνει και τόσο πολύ χρόνος για ερωταπαντήσεις, όμως θα ήθελα να απευθυνθώ στους, ε, στους συνάδελφους οι οποίοι έκαναν αυτές τις απεχθείς ε, δηλώσεις. Να τους πω λοιπόν ότι ελπίζω να μην βρεθούν ποτέ σε ανάγκη, να μην βρεθούν ποτέ σε κίνδυνο στη θάλασσα, γιατί πραγματικά... Νομίζω πως αν σας τύχει κάτι τέτοιο θα χαρείτε πάρα πολύ που υπάρχουν άνθρωποι σαν την Καρόλα Ρακέτε. Εάν περάσετε 17 μέρες πάνω σε ένα πλοίο, Νομίζω πως θα έχετε το χρόνο να διαβάσετε τον, τους νόμους και να δείτε ότι υπάρχουν ε, νόμοι οι οποίοι πραγματικά δίνουν το δικαίωμα ε, της ε, προσάραξης σε ασφαλές σε λιμάνι. Και ελπίζω λοιπόν να περάσετε 17 μέρες στη θάλασσα, να έχετε το χρόνο να καταλάβετε τι συμβαίνει. Και τα δικαστήρια είναι αυτά που θα αποφασίσουν, όχι εσείς. Και τα δικαστήρια μέχρι τώρα έχουν αποφανθεί ότι η κυρία Ρακέτα δεν είναι εγκληματίας. Αυτό ήθελα να το πω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Φέστ, έχετε ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Να απαντήσω στον κύριο Μάρκαντ. Εγώ δεν ε, έτυχε να βρεθώ σε φούσκωτο από τη Λιβύη. Δεν, έχω, δεν έχει τύχει να βρεθώ σε κίνδυνο. Κύριε Ρακέτε, υπάρχουν αναφορές ε, σύμφωνα με τις οποίες ε, Υπήρχαν, ε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ε, υπόκειται σε βασανιστήρια στην ε, Λιβύη. υπάρχουν άλλες αναφορές εφημερίδες οι οποίες λένε ότι τώρα που πήρατε αυτούς τους ανθρώπους έχουν τρεις βασανιστές λιγότερους στη Λιβύη. Σας παρακαλώ λοιπόν να μην πέφτουμε χαμηλά, να μην μιλάμε και να αποφεύγουμε να πούμε τα πράγματα με το όνομά του. Υπάρχουν τρομοκράτε, υπάρχουν βασανιστές οι οποίοι έχουν βρει το δρόμο μέσω της ε, θαλάσσιας οδού στη Μεσόγειο να αφήσουν τις ε, χώρες τους και να έρθουν στην Ευρώπη. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν εσείς είστε το χέρι που βοηθά αυτούς τους ε, τρομοκράτες και βασανιστές. Ευχαριστώ πολύ. Για ένα λεπτό, κύριε Σχοβέγγι. Ευχαριστώ πολύ. Φυσικά όλοι συμφωνούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να σώζεστε τους ανθρώπους. Είναι πολύ σημαντικό να σώσεις ανθρώπους που βρίσκονται σε κίνδυνο. Το θέμα είναι να δούμε πώς θα εξασφαλίσουμε ε, την ασφάλεια. Να μην συμβαίνει, να μην χρειάζεται να συμβεί κάτι τέτοιο. Ε, μου φάνηκε περίεργο που κάποιος από τους ευρωβουλευτές αναφέρθηκε σε νομικά δεσμευτικού κανόνε. Φυσικά και η Frontex είναι υποχρεωμένη και όλοι είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθούμε και να τηρούμε του νόμου. Όμω, τα σκάφη των μη κυβερνητικών οργανώσεων δεν θα πρέπει να είναι υπηρεσίε μεταφορά ε, προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, έτσι παραβιάζονται οι νόμοι και δημιουργείται ένα άσχημο προηγούμενο. Έτσι στέλνουμε το μήνυμα στου ε, ανθρώπου που αντιμετωπίζουν δυσκολίε στην Αφρική και αλλού ότι μπορούν να έρθουν στην Ευρώπη. Δεν θα έπρεπε να στέλνουμε τέτοιο μήνυμα. Οι μη εθνικέ οργανώσει δεν είναι ε, κράτη, δεν είναι εθνικέ αρχές και προφανώς ε, ενδέχεται να υπάρξουν και εγκληματίε σε αυτά τα ε, σκάφη που διασώζουν ανθρώπου. Ευχαριστώ πολύ. Κώστα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχάς να εκφράσω την αλληλεγγύη μου στους ε, ιδιωτικούς οργανισμούς έρευνας και διάσωσης, ε, διότι περασπίζονται τις ευρωπαϊκές αξίες, αξίες που παραβιάζουν αυτή τη στιγμή τα κράτη-μέλη και το Συμβούλιο. Η έρευνα και η διάσωση <coughs> είναι ευρωπαϊκή αξία και αυτή τη στιγμή ποινικοποιούνται και θεωρούνται εχθροί της Ευρώπης αυτοί που σώσουν ανθρώπινες ζωές. Κύριε Σότερ, μία ερώτηση σχετικά με την προσωρινή συμφωνία. Η πρόταση που έχουμε αυτή τη στιγμή αναφέρεται στα σκάφη έρευνας και διάσωσης. Τι ακριβώς ε, ε, σημαίνει αυτό και πώς ε, σκοπεύετε να κάνετε αλλαγές σε αυτό το μητρό, σε αυτό το ονειολόγιο των ε, διασωστικών πλοίων. Είναι υποχρεωμένοι να εκτελούν εντολές που θα τους δίνουν οι εθνικές συντονιστικές αρχές. Αυτές οι εντολές θα συμπεριλαμβάνουν εντολές αποβίβασης σε ασφαλή λιμάνια και θα έρχονται σε αντίθεση με το διεθνές δίκαιο ή θα συμφωνούν με το διεθνές δίκαιο της Διεθνής Συμβάσης. Ευχαριστώ κυρία Ρίβας για ένα λεπτό. Το Φεβρουάριο του 2017 στην Καταλωνία είχαμε μια πολύ μεγάλη διαδήλωση για την υποδοχή μεταναστών προσφύγων. Υπάρχει μια άλλη Ευρώπη, μια Ευρώπη που θέλει να τους καλοδεχτεί αυτούς τους ανθρώπους. Η Ισπανική κυβέρνηση ακόλουσε την πολιτική των προηγούμενων ε, κυβερνήσεων να τους στέλνει στο Μαρόκο και να στρατιωτικοποιεί τις υπηρεσίες ε, φύλαξης των ε, νότιων συνόρων. Ε, το καλοκαίρι ε, η Ισπανία κατηγόρησε την Open Arm, την απείλησε συγγνώμη, με μηνύσεις και πρόστιμα εάν συνεχίσει να διασώζει ανθρώπους στη θάλασσα. Η διάσωση στην ανοιχτή θάλασσα αναγνωρίζεται από το διεθνές δίκαιο. Δύο ερωτήσει προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι σκοπεύει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να σταματήσει αυτό το μοντέλο τη Ευρώπη Φρούριο που ποινικοποιεί την ανθρωπιστική βοήθεια και δεν τηρεί την υποχρέωσή τη για την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεύτερον, θα περάσετε πλέον στο μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Συστήματο Ασύλου να υπάρχουν νόμιμε και ασφαλεί οδοί εισόδου και να υπάρχει και ισότιμο καταμερισμό των ε, αφιχθέντων μεταξύ των κρατών μελών. Ευχαριστώ. Κύριε Ντάλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κανένας εδώ δεν είπε ότι η Λιβύη είναι ασφαλής χώρα. Εξορισμού λοιπόν, τον επιστρέφονται άνθρωποι στη Λιβύη, αναγνωρίζεται από όλου ότι είναι κατάφορη παραβίαση του νόμου από κάθε πλευρά. Δεν υπάρχει καμία αμφισημία περί αυτού. Όλοι, από όλε τι πλευρέ εδώ που αναφέρθηκαν στο κράτο δικαίου και παρόλα αυτά αυτά συμβαίνουν. Ο κύριο Λιζερή είπε ότι διασώθηκαν 2.000 ζωέ ε, στην επιχείρηση θέμη φέτο. Θα ήθελα να ξέρω πόσοι εντοπίστηκαν από τη Λιβική Ακτοφυλακή ε, από πληροφορίε που διέθεσε η Frontex. Μπορούμε να έχουμε επιβεβαίωση ότι συνέβη κάτι τέτοιο. Δόθηκαν πληροφορίε ε, για να σταματήσουν τα σκάφη και αν όντω συνέβη αυτό, τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από αυτού, τι κάνετε για να τα μεταρρυθμίσετε τη Συμφωνία του Διβλίου και αν θέλουμε να σταματήσουμε τους λαθροδιακινητέ, ε, καλύτερα θα ήταν να έχουμε ασφαλή οδό στην Ευρώπη και όχι να ποινικοποιούμε του ανθρώπου που διαθέτουν σώζουν ανθρώπους στη θάλασσα. Ευχαριστώ κύριος Λένερς. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μέχρι πολύ ενδιαφέροντα όλα τώρα μέχρι τώρα. Εγώ θα ήθελα να ξέρω τι γίνεται με αυτούς που φτάνουν ε, στις ευρωπαϊκές ακτές. Διότι δεν είναι ο ίδιος αριθμός. Το 2019 ο, η, παριθμόν ένα χώρα αφιχθέντων στην Ιταλία ήταν από την Τινησία. Και είχαμε και πάρα πολλούς ανθρώπους από το Μαρόκο. Έχουμε κάτω από 5 με 7% αναγνώριση διεθνού προστασία και για τι δύο χώρε. Ε, από νομική σκοπιά, λοιπόν, αυτό ο ορισμό ε, του ασφαλού χώρου, του place of safety, περιλαμβάνει και την διάσωση ανθρώπων στη θάλασσα από χώρε όπω το Μαρόκο και την Τινησία και δεν πρέπει αυτοί να επιστραφούν στο Μαρόκο ή στην Τινησία. Εσεί πώ αξιολογείτε την ικανότητα, για παράδειγμα, ενός πλοιάρχου, ενός εμπορικού σκάφους να αξιολογήσει αυτό το νομικό ορισμό του ασφαλούς χώρου. Και προς την κυρία Ρακέτα, Ευχαριστούμε που μοιραστήκατε την εμπειρία σας μαζί μας. Μιλήσατε για ανθρωπιστικές οδούς και νόμιμες οδούς. Δεν σημαίνει αυτό ότι όποιος θέλει να ταξιδέψει στην Ευρώπη από χώρες όπως το Μαρόκο, την Τινησία, τον Μπαγκλαντές θα πρέπει να διευκολύνεται ή θα κάνετε διάκριση εδώ μεταξύ προσφύγων που χρειάζονται διεθνή προστασία και ε, οικονομικών μεταναστών. Ευχαριστώ. Η κυρία Βόλας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ που διοργανώσατε αυτήν την ακρόαση γιατί δείχνουμε ότι δεν στρέφουμε το βλέμμα μας αλλού όταν δυσκολεύουν τα πράγματα. Είναι νομίζω πολύ εύκολα τα πράγματα. Βλέπουμε ότι έχουμε νέους ανθρώπους που κάνουν αυτό που δεν κάνουμε εμείς. Οι πολιτικοί νομίζω πως ε, πρέπει να το αναγνωρίσουν αυτό και ε, πρέπει να πάρουμε αυτό το παράδειγμα από τους ε, νέους και να αναλάβουμε τα καθήκοντά μας. Είμαστε πολιτικοί και οφείλουμε να πείσουμε και να δράσουμε. Η οδηγία για τη διευκόλυνση χρειάζεται επεξεργασία έτσι ώστε να υπάρχει με ένας διαχωρισμός ανάμεσα σε διακινητή και διασώστη. Χρειάζεται ε, επίσης να παραδεχτούμε ότι η Λιβύη δεν αποτελεί ασφαλές ε, τόπο. Χρειάζεται λοιπόν επιτέλους να πάρουμε ε, τα πράγματα στα χέρια μας και να βοηθήσουμε αυτούς ε, τους ανθρώπους μαζί με ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα να τηρούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα και εκτό επικράτεια Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμω πρέπει να γυθούμε στην προσπάθεια να ε, γίνουν κάποιε ε, κινήσεις. Τώρα, ε, όσοι έχουν διασωθεί θεωρούμε ότι θα πρέπει να παραμείνουν στην Ευρώπη. Υπάρχουν όμω άνθρωποι που βρίσκονται σε κίνδυνο, του οποίου δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε ω εγκληματίε. Υπάρχει μια κόκκινη γραμμή την οποία δεν πρέπει να ξεπεράσουμε ε, χάρη πολιτικών συμφερόντων. Σα ευχαριστώ. Ένα λεπτό παρακαλώ. Όπου να είναι θα περάσουμε μόνο στα αγγλικά. Έχετε το υπόψη σας. Έχουμε ακόμα χρόνο. Ο κύριος Ουρμπάν, για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να υπενθυμίσω μετά από τις παρεμβάσεις κάποιων από τους συναδέλφους μου εδώ στην αίθουσα που, για τις οποίες πραγματικά ντρέπομαι ότι η δημοκρατία στην Ευρώπη ε, την υπερασπίστηκε ο αντιφασισμός και σήμερα βιώνουμε πως εδώ σε αυτή τη Βουλή υπάρχουν απαντήσεις ρατσιστικές και ξενόφοβες οι οποίες και πάλι ακούγονται και αυτό είναι επονίδωστο για την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Δεύτερον, ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάρα πολύ σημαντική. Αν η Λιβύη δεν είναι ασφαλής χώρα, γιατί χρηματοδοτούμε την ακτοφυλακή της. Ποιο είναι το λιβικό κράτος, ποιον χρηματοδοτούμε, ποιον ε, καταρτίζουμε και ε, εκπαιδεύουμε στην ε, λιβική εκτοφυλακή. Νομίζω ότι είναι πολύ απλή ερώτηση. Και μία ερώτηση για τη Frontex, παρά το γεγονός ότι δεν είναι εδώ, θα ήθελα να τη στείλετε γραπτός. Συμμετού, έχετε σε έρευνα και διάσκωση στην θάλασσα του Αρβοράν. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σπούρεκ, για ένα λεπτό. Κύριε Ρακέτε, είμαι από την Πολωνία. Οπότε πρέπει να σας πω ότι εμείς είμαστε γνωστοί για την αλληλεγγύη που δείξαμε τη δεκαετία του 80. Γενναίοι άνθρωποι. Και η τρέχουσα κυβέρνηση αυτή τη στιγμή δεν δέχεται μετανάστες λέγοντας, και πρόσφυγες λέγοντας πως ας τους βοηθάμε επί τόπου. Εγώ είμαι σαφέστατα κατά αυτής της θέσης και σας ρωτώ, μια και είμαι νέα ευρωβουλευτής, τι μπορώ να κάνω εγώ, τι μπορεί να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να σας βοηθήσουμε, για να σώζετε ζωές αλλά ήδη μας είπατε στην ομιλία σας ένα κατάλογο νομοθετικών αλλαγών που πρέπει να εισάγουμε. Πείτε μας λοιπόν τι είναι το πιο σημαντικό για σας, τι μπορούμε να κάνουμε καθένας από εμά, μέσα από την καρδιά σας. Ποιο θα ήταν αυτό που θα θέλατε. Και πάλι σας ευχαριστώ για ό,τι κάνετε. Η κυρία Σάντος, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα εδώ να ε, σας καλωσορίσω